Uh, Κυρίες και κύριοι, um, λοιπόν ας ξεκινήσουμε. Ας συγκεντρώσουμε λοιπόν καταρχάς τους ομιλητές στο Προεδρείο. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμότατα στα πλαίσια της συνεδρίασης της αγοράς, εσωτερικής αγοράς, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς στα πλαίσια του Φόρουμ για την ε, ενιαία αγορά σήμερα. Είναι μια νέα προσπάθεια, πολλά υποσχόμενη. Είναι μια ιδέα η οποία περιλαμβάνεται και στην ενιαία πράξη. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Μπαρνιέ που έρχεται με τρένο στις Βρυξέλλες. Ελπίζουμε να είναι εδώ γύρω στις 3.30 ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Έχουμε εδώ και τον Βίνσεντ Βαν Κίκεμποργκ που είναι ο Ομοσπονδιακός Υπουργός υπεύθυνο για την εσωτερική αγορά. Είναι ιδιαίτερα δραστήριος στις συναντήσεις μας ο κύριος Βαν Κίκεμποργκ και μεγάλη τιμή που σας έχουμε εδώ μαζί, σας, μαζί μας. Έχουμε επίσης και τον κύριο Κόρλετς, ο οποίος είναι υφυπουργός οικονομικών στην Πολωνία. Τον βλέπω μακριά εκεί θα του δώσω το λόγο στο τέλος, γιατί μπορώ να σας ανακοινώσω επίσημα σήμερα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ένα φόρουμ πολύ πιο φιλόδοξο για την εσωτερική αγορά κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας τον Οκτώβριο του 2011 που θα κρατήσει και λίγο περισσότερο και ελπίζω να συμμετέχουν πάρα πολλοί ομιλητές από το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών και τον επιχειρηματικό κόσμο και όσους επηρεάζονται από την εσωτερική αγορά. Εμείς προσπαθούμε να εμπλακούμε περισσότερο δηλαδή από όσο μέχρι σήμερα. Ήταν μία από τις βασικές συστάσεις και της έκθεσης την οποία παρήγαγε η κοινοβουλευτική μου έκθεση. Και εδώ ένας από τους αντιπροέδρους μου, ο Λούις Γκρέκ, θα παρουσιάσει την έκθεσή του. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής έχετε στους φακέλους σας. Και επίσης μια εξαιρετική έκθεση από τον καθηγητή Μόντι, τον οποίο καλωσορίζω εδώ σήμερα. Έχετε το φάκελο, στο φάκελό σας την έκθεσή του και αυτός πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση και ενασχόληση με την εσωτερική αγορά. Με χαρά επίσης θα σας παρουσιάσω δύο πολύ σημαντικά μέλη της Επιτροπής που δούλεψαν για τα θέματα της ενιαίας αγοράς. Θα βρείτε τα ονόματά τους. Είναι η Ροζατούν από την Πολωνία και ο Κριστιαν Μπουζόη από την Ρωμανία. Βλέπετε ότι έχουμε εκπροσώπους και των σοσιαλιστών και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των φιλελευθέρων και εγώ προέρχομαι από τους συντηρητικούς Υπάρχει μια πλήρης γκάμα δηλαδή της πολιτικής. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και την παρουσία την ιδιαίτερα δραστήρια των Πρασίνων, οι οποίοι δεν είναι μένει στο Προεδρείο εδώ, αλλά συνεργάστηκαν για να φτάσουμε εδώ σήμερα. Βασική ιδέα του φόρουμ ξεκινάει από την έκθεση της κυρίας Τούνς που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον πίνακα βαθμολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήσαμε να δούμε και με άλλους τρόπους, ε, να βρούμε άλλους τρόπους να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των ε, πολιτών, όπως τα Solvit στις διάφορες χώρες. Υπάρχει μια έκθεση για τα Solvit έξω από την αίθουσα με τον Μπουζό εισηγητή. Λοιπόν, μετά από αυτή την εισαγωγή θα δώσω στους τρεις συναδέλφους μου την προεδρία της συνεδρίασης από εδώ και πέρα. Θα υπάρξει μια μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης λοιπόν από ό,τι συνήθως. Δύο-τρία πρακτικά. Δεν έχουμε χρόνο ε, για πολλές ερωτήσεις στο φόρουμ εδώ σήμερα. Τα μέλη θα κληθούν να θέσουν σύντομες ερωτήσεις στους ομιλητές μας. Σας δίνουμε επίσης την δυνατότητα να στείλετε γραπτές ερωτήσεις Έχετε ένα έγγραφο σαν γι' αυτό εδώ, ένα έντυπο σαν γι' αυτό να το συμπληρώσετε και ελπίζουμε λίγες από τις να μπορέσουμε να τις θέσουμε στους ομιλητές και να απαντήσουν. Αυτές που δεν θα απαντηθούν θα τις κρατήσουμε, θα τις κυκλοφορήσουμε και θα προσπαθήσουμε και εμείς να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, αλλά χωρίς εδώ να μπορέσω να σας εγγυηθώ το είδος των απαντήσεων. Αν πάτε στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δώσετε το όνομά σας για να σας στέλνουμε το επίσημο έντυπό μας και να γίνετε φίλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί που έχουν ενδιαφερθεί ήδη και θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται. Για να κλείσω την εισαγωγή μου. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει μία πρόταση για την ενία πράξη και ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα αναφερθεί στο θέμα αυτό όταν φτάσει. Είναι μια πρόταση η οποία έχει τεθεί προσυζήτηση για τους επόμενους τέσσερις μήνες. Υπάρχει λοιπόν η ευκαιρία η σημερινή για να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή και ο σχολιασμός. Θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Στους φακέλους σας έχετε το βαντεμέκουμ όλων των ομιλητών, δεν θα σας τους παρουσιάσω αναλυτικά θα δείτε ότι έχουμε ορισμένου πολύ διακεκριμένους ανθρώπους με πολύ συγκεκριμένο παρελθόν και ενδιαφέροντα. Είπα για τον Μάριο Μόντι, έχουμε τον Ολιβιέ Σαστέλ, τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Βελγίου που ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά και τον Φαμπιαν Τσουλάι που είναι υπεύθυνο οικονομολόγος του European Policy Center και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η κρίση στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Έχουμε επίσης και έναν πολύ έγκριτο προσκεκλημένο για τον τελευταίο γύρο μας, το τελευταίο πάνελ, Γκογέν ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο όνομα των καταναλωτών και ο Φιλίπ Ντεμπίκ, ο οποίος προσωπεί την Business Europe και με τον οποίο ενεργά συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, αυτοί θα είναι οι ομιλητές σήμερα το απόγευμα. Όσο προχωράμε θα ειδοποιούμε τους επόμενους ομιλητές. Η πρώτη ομιλία για σήμερα το απόγευμα, όπως είπα, με πολύ μεγάλη χαρά, Καλωσορίζω τον Βίνσεντ Φαν Κβίκεμπαρντ. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά με την Βελγική Προεδρία, έχουμε σημειώσει πολύ σημαντικά βήματα προόδου και αυτό οφείλεται και στη δική του εμπλοκή και αφοσίωση στα θέματα με τα οποία συνεργαζόμαστε, για τα οποία συνεργαζόμαστε. Κύριε Υπουργέ Βαν Κβίκεμπόρνε, σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Μόντι, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά μου που αποτελώ τμήμα αυτής της ε, ε, πρώτης ε, συνάντηση του Φόρουμ της Ενιά ε, Αγοράς. Η 9η Νοεμβρίου έχει γίνει πολύ συμβολική μέρα για την Ευρώπη. Ή γίνεται. Το 1988, στις 9 Νοεμβρίου, ο Ζων Μονέ, ο δημιουργός της, ε, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γεννήθηκε στη γαλλική πόλη του Κονιάκ. Το όραμά του για μια Ευρώπη ενώνει του λαού τη εξακολουθεί να ζει ακόμα και σήμερα. Και την ίδια μέρα, το 1989, γενναίοι Ευρωπαίοι κατεδάφισαν το, το τείχος του Βερολίνου αναζητώντας δημοκρατία και ειρήνη και ελευθερία. Και η ενιαία αγορά ακριβώ έχει αυτό το στόχο, να φέρει κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες και να διευρύνει τις ελευθερίες τους, να τις επεκτείνει σε όλη την Ευρώπη. Ε, το να κάνουμε την ενιαία αγορά να δουλέψει, το να την διευρύνουμε και την εμβαθύνουμε θα πρέπει να είναι ηθική μας υποχρέωση. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, ο κ. Μισελ Μπαχνιέ, έχει εργαστεί σκληρά για να συλλάβει το πνεύμα του Ζων και να το αποτυπώσει στις προτάσεις του για την ε, πράξη για την ενιαία αγορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω θεματοφύλακα των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών, έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στην λήψη των αποφάσεων σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά και η εργασία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία του Καταναλωτή, ιδιαίτερω οι συστάσεις της έκθεσης Γκρέχ, ε, είχαν ένα σαφή, ένα, σαφές, ένα σαφή αντίκτυπο στις ε, προτάσεις. Αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας την αλληγορία του Hemingway που είχε χρησιμοποιήσει ο Αλτιέρο Πινέλη παλιότερα. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τη μικρή ιστορία, το, το δίγημα του Hemingway για έναν ψαρά που αφού έπιασε το μεγαλύτερο ψάρι της ζωής του προσπάθησε να το σύρει στην, ε, στην ακτή. Αλλά σιγά σιγά καθώς έβγαινε το έτρωγαν οι καρχαρίες και όταν ο γέρος έφτασε στην ακτή το μόνο που έμενε ήταν ένα ψαροκόκαλο. Συνεπώς ε, ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε με το ίδιο πάθος ε, και την ίδια φλόγα. Και ελπίζω ότι θα καταφέρετε έτσι ώστε και το Συμβούλιο να δείξει μεγάλες ψηλές φιλοδοξίες ε, για την ε, πράξη για την νέα αγορά. Ε, μερικές ε, φορές ε, πολύ εύκολα θεωρούμε ότι έχουμε πετύχει την ενιαία αγορά, ότι έχουμε μια ενιαία, τη μεγαλύτερη αγορά των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών και των 20 εκατομμυρίων επιχειρήσεων στον κόσμο. Όμως χρειάζονται επιπλέον διαστοτικές μεταρρυθμίσεις για να αυξήσουμε την ευελιξία της, της αγορά. αγοράς. Και η έκθεση ε, παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του 2010-2011 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ε, που τη χρησιμοποίησε ως οδηγό το, συμβου... το άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας έχει εντοπίσει το μέγεθος, ε, την ελαστικότητα των αγορών μας και την ε, έλλειψη καινοτομίας, τα, τα, σημεία τα οποία καθιστούν, την, τα, οποία αποτελούν μάλλον ε, ανταγωνιστικά μειονεκτήματα της Ευρώπης σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ασία. Ε, υπάρχουν ε, τρει τομεί στου οποίου χρειάζεται δουλειά μεταρρύθμιση. Την, η αγορά των αγαθών, η αγορά των υπηρεσιών και η δημιουργία μια ενιαία ψηφιακή αγορά. Είναι τρει ε, τομεί στου οποίου αναφέρεται η πρόταση για την πράξη την ενιαία αγορά. Καταρχήν για την αγορά αγαθών. Είναι αλήθεια ότι έχουν καταργηθεί τα περισσότερα από τα εμπόδια που υπήρχαν στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών από το 1993. Η υιοθέτηση μάλιστα του πακέτου αγαθών ε, ε, δρά κίνητρο για το διασυνοριακό εμπόριο. Όμω παρόλε τις βελτιώσει, στην ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών, η προτίμηση αγορά εθνικών προϊόντων εξακολουθεί να παραμένει ψηλή. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ έχουν την τάση να ψωνίζουν τοπικά προϊόντα. Ε, ο μέσος καταναλωτής ε, ε, αγοράζει κατά 75% τοπικά ή εθνικά προϊόντα. Σε ένα βαθμό η τοπική, η εθνική προτίμηση είναι φυσιολογική. Για πολιτιστικούς ή ιστορικούς λόγους οι καταναλωτές μπορεί μάλιστα να είναι πιο απαιτητικοί σε ορισμένες χώρες από τις άλλες. Όμως σίγουρα αυτό δεν μπορεί να είναι η μόνη εξήγηση ή η εθνικη προτιμηση ειναι φυσιολογικη για πολιτιστικου η ιστορικους εξήγηση. απαιτητικοι σε ορισμενε χώρε απο τις αλλες ομως ένα άρθρο την περασμένη εβδομάδα για το Carrefour που είναι ε, το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ στην ε, Ευρώπη, που δεν μπορεί να αγοράζει τυρί ιδιωτική ετικέτα από την Ολλανδία και να το πουλάει στη Γαλλία. Και ξέρετε γιατί. Γιατί στι κάτω χώρε χρησιμοποιούν καλούπια 15 κιλών, ενώ στη Γαλλία τα τυριά, για τα τυριά χρησιμοποιούν καλούπια 40 κιλών. Συνεπώ, ε, χρειάζεται μια μεταρρύθμιση στη ρύθμιση της αγοράς των αγορών. Η Ευρώπη επίσης χρειάζεται να υιοθετήσει την έννοια της δημιουργικής καταστροφής. Χρειάζεται περισσότερους νέους καινοτόμους επιχειρηματίες και χρειάζεται καινούριε εφευρέσεις που θα διοχετευθούν στις παγκόσμιες αγορές. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που διαθέτουμε στην αγορά μας. Και τα, ε, τα παρακάτω νούμερα είναι ιδιαίτερα γλαφυρά στις 500 μεγαλύτερες ε, εταιρείες του κόσμου που ε, είχαν διαπραγματεύσει στα χρηματιστήρια, μόνο τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες δημιουργήθηκαν μετά το 1975, ενώ 26 από αυτές ε, δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ και 21 στις ε, ανερχόμενες αγορές. Ε, πρόσφατες ε, έρευνες του Ινστιτούτου Μπρούγκελ δείχνουν ότι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν εύκολα κέρδη στις όχι πλήρως ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές αγορές και αυτό τους επιτρέπει ε, να γίνουν πιο ισχυρές σε παγκόσμιες αγορές. Αυτό σημαίνει ε, ότι ε, θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα για να επιτύχει η, η πράξη για την ενιαία αγορά. Δεύτερον, ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Η ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα τα δίκτυα τηλεπικοινωνίες και τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Ε, είναι ε, σημαντική και για την ε, παραγωγή και σε άλλους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ισχυροποίηση του ανταγωνισμού σε αυτούς τους τομείς μπορεί να δώσει ωφέλη στην παραγωγικότητα και, του, πρωτογενούς, και του πρωτογενούς τομέα και στην ευημερία των πολιτών και των καταναλωτών. Ε, ο πρόεδρος, ο κύριος ε, Χάρμπορ, τόνισε στο τύπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ότι είναι πολύ σημασία να κάνουμε ε, είναι πολύ σημαντική η πρόοδος με την εισαγωγή των, σημείων, των νέων σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. η απουσία αυτόματης ή αμοιβέ αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είναι επίση ένα αδύναμο σημείο το, το οποίο τονίζει η έκθεση Μόντι οι διαφορετικές εθνικές ε, ρυθμίσεις ε, παρεμποδίζουν την δυναμική ανάπτυξη των υπηρεσιών ε, και δυσκολεύουν τους πολίτες μας να κινηθούν για να εργαστούν σε άλλες χώρες. Τρίτον, η ενιαία ψηφιακή αγορά. Έχουν γίνει πολλά ήδη για να προετοιμάσουμε την Ευρώπη για την ψηφιακή οικονομία. Η οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν ένα σημαντικό βήμα αυτό σε αυτή την πορεία. Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα ήταν το πρώτο κείμενο της Ατζέντα Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010. Αλλά και πάλι ακόμα δεν υπάρχει ενιαία ψηφιακή αγορά. Τόσο οι επιχειρήσει όσο και ο δημόσιο τομέα και οι καταναλωτέ ε, χάνουν ε, ένα τεράστιο δυναμικό ε, αύξηση της αποτελεσματικότητας της δαπάνης ε, του κάθε ευρώ τους. Κάθε κατανοητή στην Ευρώπη χάνει ε, χίλια ευρώ σε ε, αγοραστική ε, ισχύ. Και ο δημόσιος τομέας θα μπορούσε να βελτιώσει, να βελτιώσει την κατάσταση του και τα οικονομικά του με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των κρατικών υπηρεσιών. Η υπάρχει ανάγκη ε, να ε, δώσουμε ελευθερία, να απελευθερώσουμε την ενιαία αγορά ε, για τους ηλεκτρονικούς μας πολίτες. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε την προστασία των καταναλωτών, τα, τους κανόνες ευρεσιτεχνίας, να απλοποιήσουμε τους κανόνες ΦΠΑ και να εισάγουμε ψηφιακές, περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη εξουσία και δυνατότητα στον πολίτη μας ε, και να αποφύγουμε τις βλαβέρες πρακτικές. Τους επόμενους ε, μήνες ε, θα, θα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούμε προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Με την με, την καινούργια, με το καινούργιο ξεκίνημα τη ενιαία αγορά μπορούμε να ενισχύσουμε θέση των πολιτών μα και των καταναλωτών μα. Θα ήθελα να τελειώσω με κάτι που είχε πει ο Ζάμονε. Όταν μια ιδέα αντιστοιχεί στην ανάγκη της εποχής της, πάβει να ανήκει σε αυτούς που την επινόησαν. Είναι πιο ισχυρή και είναι πιο ισχυρή από αυτούς που θα την εφαρμόσουν, που θα την υλοποιήσουν. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο φόρουμ σας, το πρώτο αυτό φόρουμ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για μια ευρυτάτη παρουσίαση και για τις προκλητικές σας απόψεις για το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει καθυστερήσει ο κύριος Μόντι, λέει ο πρόεδρος. Όχι βέβαια ο κύριος Μόντι είναι εδώ, αλλά ο επίτροπος Μπαρνιέ έχει καθυστερήσει λίγο. Δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη, τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα αν δεν έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπαρνιέ. Και ο Υπουργός ε, μπορεί να δεχθεί κάποιες ερωτήσεις εφόσον εσείς το επιθυμείτε. Το λέω στους συναδέλφους μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσουν κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα, ζητώντας, ξεκινώντας τη διαδικασία από τον κύριο Υπουργό να μας ενημερώσει για ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την καινοτομία. Το δίπλωμα Ευρωπαϊκής Ευαισθητεχνίας ή το Ευρωπαϊκό μάλλον δίπλωμα Ευαισθητεχνίας έχουν γίνει πολλές συζητήσεις τον τελευταίο καιρό. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε συμφωνία. Well, thank you, um, όπως είπατε, είναι ένα από τα κεντρικά θέματα που αφορούν την καινοτομία και η ιδέα μιας ενιαίας τέτοιας, ενός, ενός τέτοιου ενιαίου διπλώματος ξεκίνησε ήδη από το 1949 από έναν γερουσιαστή Γάλλο, τον κύριο Λοσσαμπον, ο οποίος ξεκίνησε ακριβώ με την ιδέα μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ρύθμισης. Εμείς επεξεργαζόμαστε στο Συμβούλιο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόταση που ξεκίνησε ο Μπαρνιέ εδώ και λίγους μήνες, ασχολούμεθα πολύ προσεκτικά. Έχουμε οργανώσει επίσημα και ανεπίσημα συμβούλια γύρω από το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευαισθητεχνίας και θα έχουμε ένα επίσημο ε, αποφασιστικό συμβούλιο για το θέμα αύριο εδώ στις Βρυξέλλες. Και ελπίδα μας, επιθυμία μας είναι να υπάρξει συνένεση ανάμεσα στα 27 κράτη, σε όλα τα κράτη-μέλη, Οι τελευταίες 24 ώρες είναι ίσως δύσκολες. Θα εργαστώ πολύ σκληρά, όπως ακριβώς και τους τελευταίους μήνες, ημέρες και εβδομάδες, για να πείσω τους συναδέλφους μου. Νομίζω ότι στα γονίδια της βελγικής αντίληψης για τον συμβιβασμό θα βρούμε μια λύση. Μια λύση η οποία να λαμβάνει υπόψη όλες τις διαφορετικές ευαισθησίες. Είδατε ότι τους τελευταίους μήνες και σε άλλους τομείς όπως οι ρυθμίσεις για την εποπτεία, την χρηματοπιστωτική κτλ. Καταλήξαμε σε κάποιες συμφωνίες. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε την επιθυμία αυτή και πολλοί από τους εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι δεν είχαμε ποτέ φτάσει στην συνένεση από τη σήμερα τόσο κοντά. Εν πάση περιπτώσει, ας μην προκαταλάβουμε λίγο την επιτυχία, ας εργαστούμε τις τελευταίες αυτές 24 ώρες και ελπίζω αύριο κατά τη διάρκεια της νύχτας να καταλήξουμε σε μια ενιαία απόφαση. Ευχαριστώ Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που μένετε λίγο ακόμα. Ξέρω ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε τα τηλέφωνα γύρω από το θέμα αυτό σε λίγη ώρα. Έχω όμως δύο συναδέλφους που θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ πρώτη, η οποία ασχολείται με το λιανεμπόριο και Άννα Μαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ την υποστήριξή σας προς την ενιαία αγορά είναι καλοδεχούμενη. Μία πρακτική ερώτηση. Τι σκοπεύετε να κάνετε σαν Βελγική Προεδρία για να πιέσετε και να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εφαρμόσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για την εσωτερική αγορά γιατί όπως ακριβώς είπατε και δώσατε και παράδειγμα μάλιστα Υπάρχουν ε, πολλά πράγματα, όχι σε σχέση με την εφεύρεση νέων ρυθμίσεων, αλλά με την εφαρμογή των υπαρχουσών ρυθμίσεων. Καταρχά, η ε, οδηγία για τα αγαθά, η οδηγία για την λεγόμενο πίνακα βαθμολόγησης και η οδηγία για τις υπηρεσίες. Σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοθεί. Όπως είδατε στο πρόγραμμα, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Ολιβιέ Σατέλ, Σατέλ συγγνώμη, ο οποίος είναι υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα είναι σε ένα από τα επόμενα πάνελ και μια και όλοι οι καλοί Βέλγοι συνεργάζονται, μπόρεσα να, να κρυφοκοιτάξω λίγο την ομιλία του και νομίζω ότι θα σας δώσει κάποιες απαντήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ο Λιβιέ Σαστέλ θα σας δώσει την δυνατότητα και να θέσετε περαιτέρω ερωτήσεις γύρω από το θέμα που σας ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο ή μάλλον η διαφορά ανάμεσα σε ένα επιχειρηματία και τον πολιτικό είναι ότι ο πολιτικός είναι καλός στις ιδέες αλλά είναι κακός στην εκτέλεση ενώ μια γυναίκα επιχειρηματίας ή άνδρας επιχειρηματίας είναι καλύτερος σε σχέση με το εκτελεστικό κομμάτι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και νομίζω ότι ε, στο επόμενο πάνελ μπορείτε να έχετε γύρω από το θέμα αυτό μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ είναι ιδιαίτερα πετυχημένη επιχειρηματίας όπως και πολιτικός, οπότε μπορεί να τα συνδυάσει όλα. Η ιδιαιτέρως εργατική αντιπρόεδρός μου έχει το λόγο. Κοιτάξτε εδώ το ερώτημά μου αφορά περισσότερο τον Επίτροπο Μπαρνιέ, αλλά μιας και έχω το λόγο, λέει κυρία Βερνιό, κύριε Υπουργέ, σήμερα το πρωί ακούσαμε τον κύριο Λετέρνο που ήταν απεσιόδοξο σε σχέση με το δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Εσείς είσαστε λίγο πιο αισιόδοξο. Αυτό με παρηγορεί λιγάκι γιατί έχουμε να κάνουμε με μια ιδέα του Επιτρόπου Μπαρνιέ εδώ και αρκετό καιρό και σε επίπεδο κοινοβουλίου και σε επίπεδο κοινοβουλευτική επιτροπής δεν μπορούμε παρά να τον συνδράμουμε αλλά γιατί οι επιχειρήσεις, οι ερευνητέ και οι πολίτες της Ευρώπης έχουν κάθε συμφέρον έτσι ώστε αυτό το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευαισθητεχνίας που τόσο επιθυμούμε εδώ και πολύ καιρό να γίνει πραγματικότητα. Καταλαβαίνω βέβαια ότι υπάρχουν και κάποια μυστικά και κάποια επιφυλακτικότητα, αλλά πού είναι το πρόβλημα στο Συμβούλιο, γιατί εδώ διακυβεύεται το συμφέρον και του συνόλου της Ευρώπης και των μονομένων χωρών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι προσπάθειες τις οποίες έχετε κάνει η Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αξιοθαύμαστες. Και σας ευχαριστώ για αυτές. Είναι επίσης αλήθεια ότι ο Μισελ Μπαρνιέ και εγώ έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό πάρα πολύ. Έχω συναντήσει τον Μπαρνιέ πολύ περισσότερο από όσο συναντώ τη σύζυγό μου τον τελευταίο καιρό. Αλλά παρόλα αυτά για να υπάρξει μια συμφωνία απαιτείται μια πλήρη συμφωνία και μια τέτοια δεν υπάρχει. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στο θέμα που εξετάζουμε. Είναι να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό το οποίο ονομάζω σεβασμός της πολιτιστικής διαφορετικότητας, ποικιλότητα που μας κάνει δυνατούς σαν Ευρώπη και από την άλλη να βρούμε κάποια συστήματα προστασίας της καινοτομίας τα οποία να είναι συστήματα ανταγωνιστικά με αυτά που ισχύουν στη ΣΥΠΑ, στη Ιαπωνία κτλ. Το πρόβλημα λοιπόν που τίθεται είναι το τίμημα για μια μικρομεσαία επιχείρηση έτσι ώστε να καλυφθεί νομικά και να προστατεύσει ουσιαστικά το προϊόν της ε, στα εδάφη των 27 χωρών είναι κάτι το οποίο κοστίζει σήμερα 25.000 ευρώ για ένα δίπλωμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στο κόστος από τη μία, στον σεβασμό της ταυτότητας από την άλλη. Αυτό είναι το καθήκον μας και η αποστολή μας. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω ξανά τη διαπραγμάτευση στα πλαίσια αυτού του φόρουμ, καταλαβαίνετε ότι και εσείς κυρία Βερνιό έχετε μεγάλη πολιτική εμπειρία και δεν μπορώ να περάσω σε λεπτομέρειες για τις θέσεις του καθενός αλλά και ο κύριος Μπαρνιέ και εγώ ήδη σήμερα το απόγευμα το βράδυ με τη βοήθεια του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνδρομή του θα έχουμε συγκεκριμένες επαφές σε υψηλό επίπεδο και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε όλο τον κόσμο να δεχθεί αυτή τη συμβιβαστική λύση. Δεν είμαι απεσιόδοξο, δεν είμαι εκφύσεω απεσιόδοξο, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ και 35 χρόνια. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει αύριο βράδυ ένα μικρό θαύμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε πραγματικά ότι θα καταφέρετε να γράψετε ιστορία στα πλαίσια της Βελγικής Προεδρίας, ασχολούμενοι με το ζήτημα αυτό, και άλλωστε στην δική σας την πρώτη παρουσίαση αναφερθήκατε πάρα πολύ στο ζήτημα της καινοτομίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω ότι Όντω, πολλέ φορέ οι επιχειρήσει αυτέ δεν αισθάνονται αρκετά ανταγωνιστικέ σε σχέση με επιχειρήσει από άλλε πλευρέ ε, του κόσμου, σε άλλε περιοχέ του κόσμου. Σα ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ. Χαίρομαι πολύ που ο Επίτροπο Μπαρνιέ έχει πλέον φτάσει. Επομένω, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μα. Um, Δίνω αμέσω την Προεδρία στον Αντιπρόεδρο Λουίς Γκρέχ, ο οποίος θα προεδρεύσει στο επόμενο τμήμα τη συνεδρίαση Λουί. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπαρνιά, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρνιά και τον καθηγητή Μόντι που αφιερώνουν το χρόνο αυτό σήμερα και να είναι σήμερα μαζί μα. Όταν συνέταξα την έκθεσή μου όσον αφορά την πράξη ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες, φάνηκε ότι ένα βασικό εμπόδιο και σημαντική πρόκληση για την ενιαία αγορά ήταν η συμφιλίωση των αντικρουόμενων απόψεων που υπήρχαν, των τάσεων που είχαν εμφανιστεί και το πώς θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε τα διαφορετικά οικονομικά μοντέλα, προσδοκίες και προτεραιότητες των διαφόρων ενδιαφερομένων. Επίσης έγινε εμφανές ότι ήταν πολύ δύσκολο να πείσουμε ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην όλη διαδικασία να προσεγγίσουν την, το νέο έναυσμα αυτή της ενιαίας αναγοράς ακολουθώντας ε, μία πολιτική που θα επέφερε τις απαραίτητες αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υποτιμήσουμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή και θα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι τόσο ο κύριος Μπαρνιέ και ο κύριος Μόντι κατέβαλαν εξαιρετικές προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συνένεση και αυτή η συμφιλίωση. Το αν η διαδικασία αυτή θα είναι επιτυχής, αυτό εξαρτάται από όλους μας. Η, οικονομική και κοινωνική υποστήριξη όλων των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάνουμε και τη σημερινή συζήτηση. Επομένως, Καλώ αμέσω τον Επίτροπο Μπαρνιέ να πάρει το λόγο να μας παρουσιάσει την πράξη για την ενιαία αγορά και στη συνέχεια θα έχουμε 15 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Επίτροπε Μπαρνιέ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τον Λουίς Γκρέχα για την πρόσκληση, καθώς επίσης και τον πρόεδρο Μάλκομ Χάρμπορ. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου αυτή. Ήμουνα σε ένα τρένο το οποίο σταμάτησε πάνω στις ράγες για μία ώρα από κάποια άτομα τα οποία βρίσκονταν στις ράγες του τρένου. Επομένω προσπάθησα να κάνω πολύ γρήγορα προκειμένου να πάω καταρχάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία συνδυάζει αυτή τη στιγμή υπό την Προεδρία του κυρίου Μπαρόσο. Σα ευχαριστώ πολύ πάντω για την κατανόησή σα και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και που μπορώ και συμμετέχω στην πολύ μεγάλη αυτή συνεδρίαση που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είμαι εδώ παρόν μαζί σα, μαζί με όλους εσάς που με τον έναν τον άλλο τρόπο σε επίπεδο εκπροσώπηση πολιτών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων βρίσκεστε εδώ για να ακούσετε περισσότερα πράγματα για την ενιαία αγορά. Κύριε Χάρμπορ, βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο αυτής της μεγάλης δημόσιας συζήτησης για την ενιαία αγορά που θέλησε να διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα γύρω από το ζήτημα της πράξης για την ενιαία αγορά. Δεν θα αναφερθώ στους λόγους για τους οποίους βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα για να μιλήσουμε όλοι μαζί για το νέο, νέο αυτό έναυσμα που θέλουμε να δώσουμε στην ενιαία αγορά προς τους πολίτες και προς επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες. Ο καθηγητής Μάριο Μόντι που βρίσκεται δίπλα μου διαπίστωσε ξεκάθαρα στην έκθεσή του και με τις γνώσεις τις οποίες έχει το ότι υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα όσον αφορά την ενιαία αγορά, ότι συχνά δεν υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο κατανόησης, ότι πολλές φορές μάλιστα υπάρχει μία αγανάκτηση, δυσαρέσκεια από τον πολίτη καθήκον μας ως πολιτικοί, άντρες και γυναίκες, είναι να μην αρχίσουμε να αναπολούμε το παρελθόν, να μην γίνουμε νοσταλγικοί, να μην βλέπουμε επίση τα πράγματα απεσιόδοξα, αλλά να καταφέρουμε να δώσουμε μια νέα αποφασιστικότητα στο όλο εγχείρημα τη ενιαία αγορά. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάστηκα με 12 συναδέλφους υπό την αιγίδα του Προέδρου Μπαρόσο, προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε μια συνέχεια στις ε, διαπιστώσεις, στις παρατηρήσεις που κάνει στην εκθεσή του ο κύριος ε, Μόντι και προκειμένου να γίνουν κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις μετά την έκθεση την οποία συνέταξε ο Ευρωβουλευτής Λουίς Γκρέχ έκθεση την οποία μεγάλη πλειονότητα εγκρίνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι λοιπόν σε θέση να σας δώσω κάποιες πρώτες ενδείξεις πέρα από το πρώτο αυτό έγγραφο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί που αποτελεί ένα πρώτο σχέδιο της ε, ε, βίβλου αυτή η οποία θα δημοσιευθεί και που προφανώ θα μεταφραστεί σε όλε τι επίσημε γλώσσε Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία θα διοχετευθεί σε όλους τους οργανισμούς εκείνους σε επιφερειακό και εθνικό επίπεδο που επιθυμούν να συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή συζήτηση στην οποία θέλουμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν την πράξη αυτή για την ενιαία αγορά η οποία διαρθρώνεται σε τρία σημαντικά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη απέτηση των ίδιων των Ευρωπαίων και έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια ανάπτυξη πιο βιώσιμη, πιο δυνατή και πιο δίκαιη μαζί με τη συνεργασία των επιχειρήσεων. Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο λοιπόν για την ε, ανάπτυξη προσπαθήσαμε να δούμε πώς λειτουργεί η ενιαία αγορά πώς λειτουργεί ως πλατφόρμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα η νέα αγορά προκειμένου οτιδήποτε κάνουμε βασιζόμενοι σε αυτή, είτε πρόκειται για ιδιωτικέ, είτε πρόκειται για δημόσιε πρωτοβουλίε, είτε πρόκειται για εθνικέ, περιφερειακέ ή ευρωπαϊκέ πρωτοβουλίε, πώ μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα βασιζόμενε σε μια καλά λειτουργούσα πλατφόρμα. Θέλουμε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα τη ενιαίας αγορά να λειτουργεί καλύτερα και θέλουμε να πετύχουμε αυτή την επιπλέον ανάπτυξη της τάξης του 4%. Πρέπει να καταφέρουμε μαζί να πετύχουμε αυτό το 2 ή 4% επιπλέον ανάπτυξη το οποίο χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα πρέπει βέβαια να παρακολουθήσουμε στα πλαίσια της ε, ενιαίας αγοράς και τις προκλήσεις που έχουν εμφανιστεί στα πλαίσια του 21ου αιώνα. Θα εμβαθύνουμε την αγορά των υπηρεσιών βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες και θέλουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα μέσω της πολιτικής τυποποίησης. Θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα της διανομής καθώς επίσης και στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε αυτόν. Θέλουμε να καταρρύψουμε τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για ένα σύστημα ενιαίας μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ενεργειακής φορολογίας προκειμένου να γίνεται καλύτερη χρήση των ενεργειακών πόρων και να ενθαρρύνεται η χρήση των καθαρών πηγών ενέργειας. Θέλουμε επίσης κατά δεύτερο λόγο να αναφερθούμε περισσότερο στην ε, δημιουργία αυτής της νέας δημιουργικής τάσης, στις οποίες αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος Βελγικής Προεδρίας, ο Υπουργός. Και θα αναφερθώ καταρχάς στο δίπλωμα ευρεσιτεχνία. ζήτημα το οποίο με απασχόλησε ω προτεραιότητα στα πλαίσια της ε, δικής μου θητείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτημα για το οποίο βρισκόμαστε πλέον, θα έλεγα, στα τελευταία στάδια. Είναι σημαντικό λοιπόν να επικεντρωθούμε στο ζήτημα αυτό και να εκμεταλλευτούμε και τις βελτιώσεις που έχει επιφέρει η Βελγική Προεδρία. Καταλήγουμε πλέον σε μια ομοφωνία των Μάλλον πρέπει να καταλήξουμε σε ομοφωνία των ε, Υπουργών, αλλά μας μένει ακόμα δρόμος τον οποίο πρέπει να καλύψουμε. Θέλουμε επίσης ε, μια συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων του δημιουργού, καθώ επίσης και μια ενδυνάμωση τη καταπολέμησης της πειρατεία και της απομίμησης. Ξέρουμε ότι αυτές οι πρακτικέ απομίμησης καταστρέφουν 200.000 θέσει εργασία στην Ευρώπη. Τρίτο σημαντικό προσανατολισμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, που όπω το γνωρίζετε αποτελούν το 90% τη ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε λοιπόν αυτό το Small Business Act για την Ευρώπη που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Εμείς πηγαίνουμε ακόμα πιο πέρα και προτείνουμε να ενδυναμώσουμε την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, το Small Business Act, χρησιμοποιώντας την αρχή Think Small First. Να σκεφτούμε δηλαδή καταρχάς τις μικρές αυτές επιχειρήσεις, να αποτελούν αυτές προτεραιότητά μας. Θέλουμε καλύτερη πρόσβαση στα κεφάλαια για τις επιχειρήσεις αυτές. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποια περιφερειακά χρηματιστήρια και να έχουμε ειδικέ ρυθμισμένες αγορές. Επίσης να μειωθούν οι εισφορές για τις επιχειρήσεις αυτές, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει μέσω της αναθεώρησης των λογιστικών προτύπων. Τέταρτο σημαντικό προσανατολισμό, η ίδια η χρηματοδότηση τη οικονομία και η διευκόλυνση τη χρηματοδότηση αυτή. Μία βασική υποχρέωσή μου στη θέση την οποία κατέχω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να καταφέρουμε να θέσουμε τις κεφαλαγορές, τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην ε, υπηρεσία της οικονομίας, στην υπηρεσία των αγορών και όχι το αντίθετο, αυτό το οποίο έχουμε δει δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να μπορούν, να μπορούν οι αγορές αυτές να τονώσουν την οικονομία και να τονώσουν την ίδια τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη καινοτομία, περισσότερε μακροπρόθεσμε επενδύσει. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ο ίδιος αναφέρθηκε στη δημιουργία των ε, ομολόγων αυτών, κάποια ε, ομολογιακά δάνεια τα οποία θα μας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουμε ευρωπαϊκά σχέδια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων κινδύνου και θέλουμε επίσης και καλύτερες εταιρικές σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω πολλών πολιτικών οι οποίες θα προωθούν παράλληλα την ε, ενσωμάτωση, την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε και μία πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτημα των παραχωρήσεων των δημοσίων υπηρεσιών. Επίση, πρέπει να μα απασχολήσει και το ζήτημα του φορολογικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντο για τι επιχειρήσει. Όσον αφορά το φορολογικό περιβάλλον, καταρχά, έχουμε την έκθεση του Μάριου Μόντι, στα πλαίσια τη οποία προτείνεται να δημιουργηθεί μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τι επιχειρήσει και μια κοινή στρατηγική για τον φόρο προστιθέμενη αξία όπου θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα συστήματα συλλογής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Επίσης, προτείνουμε να δημιουργηθεί μια διασύνδεση των μητρών των επιχειρήσεων και να έχουμε μια αμοιβαία αναγνώριση των ε, ηλεκτρονικών συστημάτων ταυτοποίησης των επιχειρήσεων. Τέλος, κυρίες και κύριοι, Ξέρετε ότι η ενιαία αγορά στην οποία αναφερόμαστε έχει και μια εξωτερική διάσταση, μια πολύ σημαντική εξωτερική διάσταση. Μας ενδιαφέρει προφανώς ότι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και αυτό θα μας ε, απασχολήσει και στη νέα συνάντηση του G20 σύντομα θέλουμε να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ενισχύσουμε την εξωτερική μας στρατηγική βασιζόμενη σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και σε ένα πνεύμα αμοιβαίων ωφελών για όλους. Θέλουμε να προωθήσουμε περισσότερο τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προς τις τρίτες αγορές και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε την ε, μεταφορά της ε, οδηγίας για την έννοια αγορά στις συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Αναφέρομαι για παράδειγμα στις σχέσεις που έχουμε με χώρες όπως η Κίνα. Επίσης, θα ενισχυθεί η συνεργασία μας με τις τρίτες χώρες και στα πλαίσια του G20. Ένα δεύτερο σημαντικό κεφάλαιο της πράξης για την έννοια αγορά κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε και αυτοί να βρίσκονται πραγματικά στην καρδιά της ενιαίας αγοράς. Πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήθηκε ότι εξασθενεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο τις δημόσιες υπηρεσίες. Θέλουμε να αποδείξουμε εμείς το αντίθετο και θέλουμε να δείξουμε ότι όντως οι υπηρεσίες αυτές μπορούν πραγματικά, μάλλον οι, Ευρω ευρωπαϊκοί κανόνε και τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα μπορούν να υποστηρίξουν τι δημόσιε υπηρεσίε σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο το 2011 θα προτείνουμε ε, νέε προτάσει όσον αφορά τι υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο. Πρόκειται για δέσμευση του Προέδρου Παρόσο και γι' αυτό το λόγο προτείνεται μία δέσμη μέτρων προς τις δημόσιες υπηρεσίες για να έχουμε μία καλύτερη αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους τους χρήστες, μία αξιολόγηση των καθολικών υπηρεσιών που θα πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να αποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών. Ο συνάδελφός μου κύριος Αλμούνια θα εξετάσει επίσης τη δέσμη Monty Cross, το πακέτο αυτό μέτρων που έχει να κάνει με την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης θα κάνουμε κάποιες προτάσεις για να βελτιωθεί το δίκτυο υποδομής. Πρόκειται δηλαδή για κάποιες ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες. Θα δώσουμε νέους προσανατολισμούς όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών. Θα αναφερθούμε στο σφαιρικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των υποδομών αυτών και θα δώσουμε μέχρι το 2020 ιδιαίτερα έμφαση στα ενεργειακά δίκτυα και θέλουμε να ενσωματώσουμε σε αυτά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο δεύτερο αυτό κεφάλαιο υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο που έχει να κάνει με την αλληλεγγύη. Πολύ συχνά η κοινή γνώμη θεωρεί ότι ε, η ενιαία αγορά θέτει ένα αμφιβόλο τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Τα πρόψή μου ξεκάθαρα με τις συνθήκες της Λισαβόνας και με τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων η νομοθεσία της ενιαίας αγοράς σε καμία περίπτωση δεν θέτει εμπόδια στην ε, δυνατότητα συλλογικών ε, προσφυγών. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε μια οριζόντια κοινωνική ρήτρα σε όλα τα νομεθήμετά μας όπως το απαιτεί αυτό και η συνθήκη της Λισαβόνας. Τι προτείνουμε λοιπόν γι' αυτό. Και γι' αυτό βέβαια θέλουμε και τη δική σας συμβολή. Θέλουμε να έχουμε μία συστηματική αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων όλων των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων να αξιολογήσουμε καλύτερα την ε, οδηγία που έχει να κάνει με την απόσπαση των εργαζομένων και να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά για την ε, καταπολέμηση της παράκαμψης των ε, κανόνων. Θέλουμε επίσης να έχουμε έναν πραγματικό κοινωνικό διάλογο στις εργασιακές σχέσεις. Τρίτον, στα πλαίσια πάντα της αλληλεγγύης, Θέλουμε ο καθένα στα πλαίσια τη ζωή του να μπορεί να υποφελείται τη ενιαία αγορά και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε κάποια μέτρα για την πρόσβαση σε θέσει απασχόληση καθώ επίση και σε καλύτερα προγράμματα κατάρτιση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα καθώ επίση και καλύτερα μια εναρμόνιση των συστημάτων, εθνικών συστημάτων κατάρτιση. Τέταρτη δέσμη μέτρων. Αναφέρθηκα στην ανταγωνιστικότητα ήδη από την αρχή τη παρουσίασή μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνοδευτούν τα μέτρα αυτά από κάποια νέα μέσα για να προωθηθεί η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Θέλουμε εδώ πέρα να έχουμε μεγαλύτερη κοινωνική επιχειρηματικότητα και θέλουμε να βελτιώσουμε το νομικό πλαίσιο των επιχειρήσεων εκείνων που καινοτομούν κοινωνικά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, μία σήμανση για αυτές τις κοινωνικά υπεύθυνε επιχειρήσεις και θέλουμε μία καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών σε μέσα χρηματοδότησης. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε, για παράδειγμα, τις επενδύσεις ή μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο επενδύσεων το οποίο θα μπορούσε χρηματοδοτικά να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις αυτές. Προτείνουμε επίσης μία αναδιάρθρωση της διαχείρισης των επιχειρήσεων προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτές οι οποίες είναι πιο κοινωνικά υπεύθυνες. Πέμπτον, θέλουμε να καταστήσουμε την ενιαία αγορά πιο προσβάσιμη για όλους τους καταναλωτές σε πολλούς τομείς. Όσον αφορά την γενικότερη ασφάλεια των προϊόντων, καλύτερη πληροφόρηση, και καλύτερη προστασία των καταναλωτών, ιδίως για τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες, με μια συγκεκριμένη οδηγία για την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές τραπεζικές υπηρεσίες βάσης, καθώς επίσης και στα ενυπόθηκα δάνεια. Θέλουμε να καταρρύψουμε όλα τα φορολογικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν για του πολίτε κάθε φορά που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά και θέλουμε επίση να δυναμώσουμε τα δικαιώματα των επιβατών σε κάθε μέθοδο κυκλοφορία και μετάβαση για όλου του τρόπου μεταφορών. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να περάσω στο τρίτο τμήμα, στο τρίτο σημαντικό κεφάλαιο της πράξης για την ενιαία αγορά και να αναφερθώ περισσότερο εδώ πέρα στον διάλογο και στην εταιρική σχέση. Αναφερθήκατε κύριε Πρόεδρε και εσεί ο ίδιος στη νέα αυτή σημαντική μέθοδο την οποία έχουμε, δηλαδή την διαβούλευση τον διάλογο, θα ήθελα πολύ γρήγορα να αφαιρθώ σε κάποιες προτεραιότητες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο σε μια ευφυή ρύθμιση, ευφυή νομοθεσία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενδυναμωμένη συνεργασία όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε περισσότερο διάλογο και καλύτερε προτάσει. Θέλουμε έπειτα καλύτερη μεταφορά και εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Και πάλι εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μια καλή εταιρική σχέση και ένα διάλογο με τα κράτη-μέλη και μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε παντού το σύστημα Solvit, το οποίο λειτουργεί παντού. Τρίτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία θηρίδα πληροφόρηση, καθώ επίση και μια ενιαία θηρίδα προσφυγή των πολιτών, προκειμένου να καταφέρουμε να βρίσκουμε εξώδικε λύσει σε προβλήματα που προκύπτουν. Τέλο, θέλουμε εταιρική σχέση και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Στην ουσία, θέλουμε εδώ πέρα να έχουμε ένα κατάλογο top 20, δηλαδή των σημαντικών ετοιμάτων που έχουν οι σημαντικοί παράγοντες στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς και θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε σε αιτήσια βάση και αυτό το φόρουμ αγοράς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε πάντα να αξιολογούμε την πρόοδο που επιτυχάνεται ή να καταφέρουμε να ελέγχουμε τα εμπόδια τα οποία προκύπτουν. Εν κατακλείδη κύριε Πρόεδρε, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στον διάλογο Έμπρακτη απόδειξη του διαλόγου αυτού είναι η σημαντική σημερινή συνεδρίαση. Η πράξη για την ενιαία αγορά δεν είναι ασύνηθε έγγραφο. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράση, το οποίο με συλλογικό τρόπο επεξεργαστήκαμε με 12 συναδέλφου μου. Είναι ένα έγγραφο το οποίο περιέχει 50 προτάσει. Όλε θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες, ορισμένε περισσότερο από τι άλλε, Κατά τη διάρκεια συζήτηση θα δούμε ποιε είναι ε, οι προτάσει προτεραιότητα ενδεχομένω να πρέπει ορισμένε από τι προτάσει αυτέ να ενδυναμωθούν, ενδεχομένω να πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποιε άλλε, ενδεχομένω να έχουμε κάνει και πάρα πολλέ προτάσει, ενδεχομένω να πρέπει να τι μειώσουμε. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε ακριβώ το διάλογο αυτό, ξεκινώντα από τι 50 αυτέ προτάσει και θέλουμε κατά τη διάρκεια τη ε, συζήτηση αυτή ε, να είμαστε πραγματικά και εγώ και οι συναδελφοί μου πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία θα μα πείτε. Σας το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια. Σας προτείνω λοιπόν να κλείσουμε τον κατάλογο προτεραιοτήτων σε αυτές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και ελπίζουμε κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012 να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τις προτάσεις αυτές. Κατά αυτόν τον τρόπο, την 20η επέτειο της ενιαίας αγοράς θα είμαστε σε θέση να μην είμαστε μελαγχολικοί, νοσταλγικοί, αλλά αντίθετα θα είμαστε σε θέση να δείξουμε δυναμικότητα, βούληση, ακριβώς αυτά τα οποία περιμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες σε μια περίοδο ανησυχία, σε μια περίοδο που ακόμα διανύουμε μια σημαντική οικονομική κρίση. Μια περίοδο η οποία θα μας επιτρέψει να αντλήσουμε τα κατάλληλα διδάγματα διδάγματα τα οποία θα μας επιτρέψουμε, να, να, θα μας επιτρέψουμε συγχωρείτε, να έχουμε μια πιο προληπτική στάση, μια πιο προδραστική νομοθεσία. Προσπάθησα σύντομα να σας περιγράψω το περιεχόμενο αυτής της πράξης για την ενιαία αγορά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας στις Βρυξέλλες και σε όλα τα κράτη-μέλη για να συμμετέχω σε, μια, σε ένα δυναμικό διάλογο προκειμένου να δώσουμε νέα όθηση για την ενιαία αγορά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όλοι όσοι θέσουν ερωτήσεις παρακαλώ να περιοριστούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και Σφάπ. Κύριε Σφάπ, έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον Επιτρόπο Μπαρνιέ για τον τίτλο της ανακοίνωσης του. υπέρ μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς εξόχου ε, εξόχους ανταγωνιστικής. Εξαιρετικός ο τίτλος, είναι πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική πρόοδος. Αυτό που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα είναι να εξετάσουμε πώς θα δώσουμε καλύτερο προσανατολισμό στην ε, εσωτερική αγορά τα επόμενα χρόνια. Η πρόταση της ε, Κομισιόν αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και μια εξαιρετική πρώτη τοποθέτηση. Βέβαια χρειάζεται να εμβαθύνουμε σε αυτές τις ιδέες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την φάση της διαβούλευσης. Πολύ καλό να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πριν ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη μεριά του θα συμμετάσχει όσο πιο δραστηρία γίνεται και ιδιαίτερως η Επιτροπή μας. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας πιστεύω ότι η ενιαία εσωτερική αγορά θα προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ που συμπεριλάβατε και τα, ε, στην έκθεση σας. Πολύ ωραία. Ε, η κυρία Βερνιό. Οι συντονιστέ ήταν να μιλήσουν πρώτοι, έτσι είχαμε συμφωνήσει. Εν πάση περιπτώσει, με ξέπληξε που μου δώσατε το λόγο, Εμπερναντέτ, θα το κάνει εξίσου καλά. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μπαρνιέ, συγχαρητήρια. Ε, τα περισσότερα από όσα συμπεριλέβαν ο κ. Μόντ και ο κ. Γκρέξ στι εκθέσει του, ε, τα έχετε και εσεί συμπεριλάβει στην ανακοίνωσή σα. Ιδιαίτερα αυτή η σφαιρική προσέγγιση που ακολουθείτε είναι πάρα πολύ καλή. Όμω, δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στην κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο συμφέρον των εταιριών και το συμφέρον των πολιτών μας. Είμαστε πολύ μακριά από αυτήν την ισορροπία μάλιστα θα έλεγα. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες αλλά θα εστιαστώ σε τρία σημεία. Η ομάδα μου υποστηρίζει παγίως ότι χρειαζόμαστε ε, μια χρειαζόμαστε κοινωνικούς στόχους στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Δηλαδή, η κοινωνική συνιστόσα είναι σημαντικό κομμάτι της πολιτικής δουλειάς μας. Αυτό όμως έχει υποβαθμιστεί πολύ στις μελέτες, έχει πάρει τη μορφή μελέτης αντικτύπου μόνο πλέον. Δεύτερον, συζητούμε εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια το θέμα των συλλογικών προσφυγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει άπειρε μελέτε, έχει εκδώσει εκθέσει και τελικά τι βλέπω στι προτάσει σα, ότι χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερε μελέτε. Δεν κάνετε προτάσει για το πώ θα εφαρμοστεί αυτό. Αδυναμία. Αδυναμία και κενό κρίμα που δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο εκεί. Τρίτο, σημείο τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες ενδιαφερόμαστε εμείς ως ε, σοσιαλιστές δημοκράτες. Ε, δεν το αντιμετωπίζετε σωστά στην εκθέση σας. Χρειαζόμαστε μια, ένα πλαίσιο προστασίας αυτών των υπηρεσιών καθολικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Εγώ ξέρω ότι έχετε τη βούληση να προχωρήσετε σε αυτό το θέμα και σας προσφέρουμε τη συνεργασία μας. Θα κάνουμε και προτάσεις. Ευχαριστώ. Thank you. We pass it on to the coordinators first. Πρώτα οι συντονιστές, ε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, έχετε υποβάλει 50 προτάσεις για την ενιαία εσωτερική αγορά. Πολλές από αυτές είναι πολύ ειδικέ και αυτό είναι καλό. Κάποιες δεν είναι πολύ θετικές ή είναι πολύ γενικέ. Για παράδειγμα, σα σας δώσω ένα παράδειγμα, ψηφιακή αγορά. Ο καθηγητής Μοντή έχει αναφέρει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Χρειάζεται να αποκτήσουμε ένα πλαίσιο. Πλαίσιο έτσι ώστε οι υπηρεσίες να αποκτήσουν ένα ελκυστικό περιεχόμενο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Κάτι που δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Μια άλλη αδυναμία πολλές παρανομίες γίνονται στον ψηφιακό κόσμο. Είναι περίπλοκο και αδιαφανές το πλαίσιο λειτουργίας τους και παροχής αυτών των υπηρεσιών και χρειάζεται να το διευκρινίσουμε, να το απλοποιήσουμε προς όφελος και των καλλιτεχνών και των καταναλωτών. Γιατί αλλιώς ποιος θα μας πάρει στα σοβαρά. Λοιπόν, ας είμαστε πιο φιλόδοξοι, ιδιαίτερα στο θέμα της ψηφιακής αγοράς. Σε πολλές από τις προτάσεις σας συμφωνούμε ως Κοινοβούλιο. Είναι πολύ θετικές, είναι πολύ καλές. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την νέα εσωτερικορά και να την προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Κυρία Ρούλε, θα ήθελα να περιστώ σε δύο σημεία. Συμφωνώ με την κυρία Γκέφαρτ σε πολλά σημεία, σε πολλά από αυτά που είπε για το θέμα υπράγματος συλλογικών προσφυγών. Όμω, έχω και κάποια άλλα πράγματα. Είπατε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε θέματα φορολόγηση και ιδιαίτερα στη φορολόγηση της πράσινης ενέργειας. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσατε όμως να ε, δώσετε λίγο περισσότερο βάρος στις προτάσεις σα στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί δεν αναφέρεται καθόλου η κλιματική αλλαγή και πολλά άλλα πράγματα. Θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο αυτέ τι προτάσει σα. Δηλαδή αν είχαμε μια ανάπτυξη 3-4% βιώσιμη θα ήταν καλά. Αλλά αν όμω αυτή η ανάπτυξη γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος και εντείνει τις κλιματικές αλλαγές, ε, δεν είναι θετική ε, καλή ανάπτυξη. Μετά η διαφάνεια, πολύ σημαντική, είπατε ότι θα ανοίξουν οι ομάδες των προγνωμόνων. Ε, εμείς ως κοινοβούλιο ασφαλώς και θα συμφωνήσουμε στο να είμαστε περισσότερο ε, ενημερωμένοι για την εργασία που κάνουν οι προγνωμόνες στην Κομισιόν ιδιαίτερα αν γνωρίζαμε τη σύσταση των ομάδων πυρογνωμόνων. Σίγουρα πολύ θετικό. Το άλλο πράγμα που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις ε, σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς οι πολίτες θα πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο, να μπορούν να πούν τη γνώμη τους και να εισακουστούν. Και επανέρχομαι στο πώς γίνονται οι ακροάσεις στην Κομισιόν. Δεν γίνονται με αρκετά διαφανή τρόπο και δεν γνωρίζουμε τι συμπεράσματα βγαίνουν από τις ακροάσεις που κάνει η Κομισιόν. Ένα παράδειγμα. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλές ε, απόψεις για τις εκχωρήσεις ε, και γίνονται ακροάσει, ε, πολλοί εκφράζουν την άποψή του και τελικά ε, η Κομισιόν δεν τι λαμβάνει υπόψη. Πολλοί αναρωτιόνται γιατί συμμετέχουν στι ε, ακροάσει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια, να ξέρουμε ποιο πρότεινε τι και τι πρότεινε η πλειοψηφία, εν περιπτώσει, για να ξέρουμε αν ακολουθήθηκε η γνώμη τη ή όχι. Αυτό το οφείλουμε στους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ο κ. Τριανταφυλλίδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναφορικά με τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος για τις οποίες μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι προηγουμένως, αναφερθήκατε στην επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας τους. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να δώσετε λίγα περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό το σημείο, δηλαδή προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αλλαγή του χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών. Λέγοντας χαρακτήρα, η ανησυχία μου είναι αυτές οι υπηρεσίες να μετεξελιχθούν από υπηρεσίες για όλους σε υπηρεσίες για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να τις αποκτήσουν. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπανιέ για να απαντήσει. Θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις. Καταρχάς ευχαριστώ τους συντονιστές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και λυπάμαι που θα φύγω αμέσως μετά. Αλλά θα αφήσω τα αυτιά μου στην αίθουσα και θα μου πούν το τι θα πείτε, τι προτάσεις θα κάνετε και τι επικοδομητικές κριτικές θα σημειώσουμε γιατί πρέπει να πάω στη συνεδρίαση του συνόλου των επιτρόπων αργότερα. Ευχαριστώ τον κύριο Σφάμπ, γιατί έδειξε ότι κατάλαβε πολύ καλά ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι η ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς να γίνει στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Και οι τρεις λέξεις έχουν σημασία. Και θα μπορούσα να προσθέσω και το ιδιαίτερο ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, γιατί αυτό λέει η συνθήκη. Όλες οι λέξεις έχουν σημασία οικονομία, κοινωνική οικονομία της αγοράς και καμία από τις λέξεις αυτές δεν είναι ύβρις. Για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, για να ξαναβρούμε, να ξανασυναντήσουμε την ανταγωνιστικότητα, να την ανακτήσουμε, θα πρέπει να πούμε ότι όλοι είμαστε απαραίτητοι. Κάθε πολίτης είναι απαραίτητος, κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητη, κάθε ομαδοποίηση δημοτική, κοινοτική αν θέλετε είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε να πετύχουμε χωρίς τον τεράστιο αριθμό των μικρομεσαίων σαν παράδειγμα στην Ευρώπη. Η επόμενη συνάδελφος αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα που αποτελούν τις ανησυχίες της πολιτικής της ομάδας. Θα κάνουμε και εμείς προτάσεις για τη δράση μας και συλλογικά η κυρία Ρέντινγκ και ο κύριος Σαλμούνια. Περιμένω επίσης και τις, περιμένω μάλλον κατανοώ τις προσδοκίες σας σχετικά με την κοινωνική ρήτρα χωρίς να προδώσω τίποτα. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το θέμα είχαμε σε βάθος συζητήσει στο σύνολο των Επιτρόπων και το κείμενο το οποίο είναι υποσυζήτηση είναι ένα κείμενο που ισορροπεί θα έλεγα διαφορετικές ευαισθησίες που πρέπει να εκφραστούν όλες. Και στο θέμα αυτό και στα υπόλοιπα θέματα στα οποία εμένω εγώ όπως το θέμα της απλούστευσης των εγγυήσεων για την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινή ωφέλεια υψηλή ποιότητα. Ξεκινάμε τη συζήτηση εκ νέου γιατί θέλουμε να υπηρετήσουμε σωστά όλων τις προσδοκίες, θεμητές προσδοκίες που εκφράζονται από όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν αναφέρθηκα στην ομιλία μου τη σύντομη στο σύνολο των προβλημάτων, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία συνεργάζομαι με την Ελικρός, την εμβάθυνση σαν παράδειγμα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Αυτό αφορά επίσης και το δικαίωμα ευαισθητεχνίας, είναι κάτι στο οποίο εμένω ιδιαιτέρως. Αλλά θα ήθελα να εξυγχρονιστεί το σύστημα στα πλαίσια του διαδικτύου, να προστατεύονται οι εφευρέσεις φυσικά και στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου που δεν αντιπροσωπεύει βέβαια ακόμα παρά μόνο το 2% των εμπορικών συναλλαγών. Την ψηφιακή υπογραφή, το ψηφιακό εμπόριο γενικότερα, πολλά μένει να γίνουν για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Για την κυρία Ρουλέ. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρανοήσεις και το λέω επανειλημμένα δεν φιλοδοξούμε να καλύψουμε όλα τα πολιτικά προβλήματα και όλες τις στρατηγικές. Λέω συχνά ότι η ενιαία αγορά είναι η βάση της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι η πλατφόρμα. Πάνω σε αυτήν εδράζεται η οικονομική δραστηριότητα. Πάνω σε αυτήν την αγορά, πάνω σε αυτήν την ενιαία αγορά θα οικοδομήσουμε τη στρατηγική μας. Κυρία ρουλέ, έχουμε διαφορές σε κάποια θέματα, διαφορετικές απόψεις. Αλλά η νέα μορφή ανάπτυξης την οποία επιδιώκουμε θα πρέπει να είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Δεν θα παραμείνουμε στα ίδια και σε επίπεδο διακανονισμών ρυθμίσεων και σε επίπεδο εποπτείας. Δεν περιοριζόμαστε στην αυτορύθμιση της αγοράς. Η διακυβέρνηση της αγοράς είναι μια νέα ευθύνη και η ανάπτυξη που θα οικοδομήσουμε θα είναι αλλιώτικη αυτή τη φορά. Θα είναι δίκαιη, θα είναι ποιοτικότερη, λαμβάνοντας υπόψη το ότι οι φυσικοί πόροι και ο φυσικός χώρος δεν είναι πλέον δωρεάν για κανέναν και δεν είναι τίποτα πλέον ανεξάντλητο και δωρεάν. Αυτό πρέπει να το ε, σημειώσουμε για το καλό το δικό μας και των επομένων γενεών. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτή της ενίας πράξης, όλες οι στρατηγικές που ακολουθούμε για την αηφορία <clears throat> δεν μπορεί παρά να ληφθούν υπόψη. Για τις ε, παραχωρήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, Νομίζω ότι έχουμε δίκιο να προχωρήσουμε σε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν έχουμε ακόμα τις τελικές προτάσεις. Περιμένουμε το τέλος των διαπραγματεύσεων για να καταλήξω σε ορισμένες προτάσεις οι οποίες ελπίζω να είναι πραγματιστικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, κάποιες, ε, κάποιοι κανόνες, κάποιο πλαίσιο ρυθμιστικό βέβαιο νομικά για τις εκχωρήσεις ιδιαίτερα στον τομέα των υποχρεώσεων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε προβλήματα στις τοπικές αρχές ε, για τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Όπως και η κυρία Γκέπχαρτ αναφέρθηκε στις υπηρεσίες καθολικού συμφέροντος. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια σε βάθος συζήτηση. Έχουμε προχωρήσει σε διευκρίνηση των προβλημάτων. Έχουμε ορίσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα και των κρατικών επιχορηγήσεων και βοηθειών. Είμαστε έτοιμοι για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εδώ είναι το σημερινό πλαίσιο, εδώ βρισκόμαστε. Θα πρέπει να μας πείτε κι εσείς, σαν κοινοβούλιο, θα πρέπει να μας πούν και τα εθνικά κοινοβούλια, θα πρέπει να μας πούν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Εγώ έχω αναλάβει την υποχρέωση να ακούσω τις προτάσεις σας και να μην προτείνω τίποτα σαν υπεύθυνο για την εσωτερική αγορά που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τον κάθε πολίτη, ιδιαίτερα τον πιο εύθραστο πολίτη, τον πιο απομονωμένο πολίτη από την πρόσβασή του την ανεμπόδιστη σε υπηρεσίες καθολικού συμφέροντος υψηλής ποιότητας. Όπως είχε συστήσει ο Γκρέσ και ο Μάριο Μόντι, εγώ προσπάθησα να παρουσιάσω μια σφαιρική άποψη και πρέπει να φύγω τώρα για την εσωτερική αγορά. Προσπάθησα να καλύψω αρκετές ανησυχίες με συγκεκριμένο τρόπο, αρκετές φοβίες και αρκετά ε, ερωτηματικά τα οποία δημιουργεί ένας λαϊκισμός και ένας κάποιος προστατευτισμός. Το πρώτο θύμα του προστατευτισμού θα είναι η εσωτερική αγορά για να καταπολεμήσουμε αυτές, αυτούς τους πειρασμούς τους λαϊκιστικούς και τους προστατευτικούς νομίζω χρειαζόμαστε νέες προτάσεις. Κάναμε 50 νέες τέτοιες προτάσεις. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίες, είναι πραγματιστικές, είναι προοδευτικές ε, θα σας ακούσουμε προσεκτικά τον επόμενο Φλεβάρι θα μας κάνετε τις προτάσεις σας και πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών θα συνεισφέρουν στη συζήτηση και θα στηρίξουν το πρόγραμμα ανάκαμψης της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέρα από αυτή τη σύντομη παρουσία μου εδώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Δυστυχώς δεν έχουμε. χρόνο για περισσότερες ερωτήσεις. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπαρνιέ και θα ακούσουμε τον κύριο Μόντι. Now I request Professor Monti, who's Δίνω το λόγο στον κύριο Μόντι, πολύ σημαντικό πρωταγωνιστή και παράγοντα για την ενιαία αγορά, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να δώσουμε, να προκαλέσουμε αυτή την ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα το ότι μπορώ και συμμετέχω σε αυτό το φόρουμ ενιαίας αγοράς και ήταν ιδιαίτερα εγκαρδιωτικά τα όσα άκουσα από τον κύριο Χάρμπορ, από τον Υπουργό και από τον Επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος έκανε μια παρουσίαση της πράξης για την έννοια αγορά. Κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ πολύ για την διοργάνωση της ε, σημερινής συζήτησης και νομίζω ότι ο διάλογος αυτός αποτελεί πολύ σημαντικό πυλώνα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Βλέπουμε ένα καταπληκτικό παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα συμβαλόμενα μέρη τα οποία βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους ιδιαίτερος τον ε, Μισελ Μπαρνιέ για την πράξη για την ενιαία αγορά. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε έναν άνθρωπο με τέτοια εμπειρία, αποφασιστικότητα, αφοσίωση στο ευρωπαϊκό ιδεώδες, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ηγέτης της νέας αυτής προσπάθειας για την καθίδρυση της πράξης για την ενιαία αγορά. Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση την οποία περιέγραψε ο Επίτροπος Μπαρνιέ και στην ε, έκθεση την οποία υπέβαλα εγώ μετά από αίτημα του Πρόεδρου Μπαρόσο υπάρχει και ένα κεφάλαιο το οποίο τυπλοφορείται μία ενιαία αγορά για την επίτευξη ενός ανώτατου επίπεδου ανταγωνισμού, ανταγωνιστικότητας, με συγχωρείτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί όντω ένα πολύ σημαντικό κριτήριο συγκριτική αξιολόγηση για τι μελλοντικέ προτάσει. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ στη δική του πρόταση για μια πράξη για την ενιαία αγορά προτείνει να γίνει κάτι το οποίο δεν είχε αρχικά πριν από ένα χρόνο γνωριστεί ως προτεραιότητα, ως αναγκαιότητα. Δηλαδή, να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των πολιτών και οι κοινωνικές ανησυχίες ως αναπόσπαστο τμήμα της προσπάθειας, το οποίο αν δεν ληφθεί υπόψη θα εμποδίσει την περαιτέρω εξέλιξη της ενιαίας αγοράς ή μπορεί ακόμα και να μας γυρίσει πίσω σε περιόδους οικονομικού προστατευτισμού. Θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ για να ενισχυθεί περισσότερο η όλη συζήτηση που ξεκινάει σήμερα. Να σας πω ότι μου προκάλεσε εντύπωση το ότι είδα ότι προβλέπεται μία τετράμινη περίοδος διαβούλευσης και συζήτησης και μου προκάλεσε αυτό εντύπωση γιατί θεωρώ ότι ε, το να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην νέα αγορά είναι κάτι το ιδιαίτερα επίγον. Κάτι το ιδιαίτερα επίγον, ιδίως όσον αφορά την ε, λήψη αποφάσεων και ιδίω να λάβουμε υπόψη την όλη διαδικασία λήψη αποφάσεων που είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα χρονοβόρα και ιδίω να λάβουμε υπόψη μας και την οικονομική κρίση την οποία διανύουμε. Θεώρησα λοιπόν ότι η πράξη για την ενιαία αγορά θα μπορούσε λίγο πιο άμεσα να μας βοηθήσει να λάβουμε τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε. Εκ μέρους ε, του Πρόεδρου Μπαρόσο αφιέρωσα έξι μήνες για διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και με όλους, του τους ενδιαφερομένους. Και οι ευρωβουλευτές γνωρίζουν, φαντάζομαι, ότι οι διαβουλεύσεις αυτές γίνανε με κάθε ένα και το υπογραμμίζω με κάθε μία από τις πολιτικές σας ομάδες και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ξεκινώντας από την Επιτροπή εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς είχε και το σύνηθες πάνελ ενδιαφερομένων, το οποίο και αυτό συνεδρίασε. Επίσης, κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να γίνουν και διαβουλεύσεις για συγκεκριμένα νομοθετήματα, για συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Και αυτό θα γίνει βέβαια υπό το πνεύμα της έκθεσης του Λουίς Γκρέχ. Δηλαδή θα έχουμε συγκεκριμένα φόρα κάθε φορά, τα οποία θα ασχολούνται με επιμέρους νομοθετήματα. Επομένω, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πραγματικά χρειάζονται αυτοί οι τέσσερις μήνες δημόσια συζήτησης. Επίσης πιστεύω ότι η ενιαία αγορά υποφέρει όχι τόσο από την απουσία διαβουλεύσεων για το τι θα πρέπει να γίνει, υποφέρει μάλλον από την απουσία πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δαχοκοκαλιά της ε, έκθεσής μου είναι το εξής ερώτημα. Από πού θα έρθει η πολιτική ενέργεια. Η άποψή μου είναι ότι η πολιτική αυτή ενέργεια δεν θα έρθει μέσα από συνεχιζόμενους κύκλους διαπραγματεύσεων. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Σαφώς είναι χρήσιμες οι διαβουλεύσεις, αλλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να καινοτομήσουμε κατά κάποιο τρόπο, να καταφέρουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν αντικρουόμενες απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα να συμφωνήσουν. Και γι' αυτό το λόγο η έκθεση που υπέβαλα για τον πρόεδρο Μπαρόσο προσπαθεί να εντοπίσει τα σημεία εκείνα στα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί μια κάποια συμφωνία. Προσπαθώ να βρω δηλαδή κάποιους ε, τομεί όπου θα μπορούσε να υπάρχει συνένεση ανάμεσα σε κράτη-μέλη τα οποία προωθούν περισσότερο μια ελεύθερη προσέγγιση της αγοράς και σε κράτη-μέλη που έχουν μια πιο κοινωνική προσέγγιση της αγοράς. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν φέροντας την νέα αγορά στο κέντρο της πολιτικής προσοχής. Ο κύριος Γκρές το γνωρίζει και πολλά μέλη επίση του Κοινοβουλίου ότι σε πολλέ συζητήσει που είχαμε μαζί είδαμε ότι το πρόβλημα τη ενίσχυση αγορά δεν είναι μόνο η δυσκολία αυτή καθ' αυτή που παρουσιάζει, αλλά το ότι δεν καταφέρνει να κεντρήσει την προσοχή κάποιων πολύ σημαντικών πολιτικών παραγόντων στην Ευρώπη. Δεν βρίσκεται δηλαδή στο κέντρο τη πολιτική συζήτηση, των πολιτικών προτεραιοτήτων. Για άλλη μια φορά όμω δεν επετεύχθη αυτό μετά την υποβολή τη πρόταση για την πράξη για την ενιαία αγορά. Εγώ αυτό ήλπιζα στην αρχή. Ήλπιζα ότι το ζήτημα αυτό θα έπαιρνε ιδιαίτερη κάλυψη στα μέσα μαζική ενημέρωση. Ότι κάπου θα διαβάζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει μια πολύ γενναία θαραλέα πρωτοβουλία. Δυστυχώ δεν είδαμε κάτι τέτοιο ακόμα και η μικρή, κάποια παραμικρή απόφαση για ρύθμιση για παράδειγμα των hedge funds λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ότι η ίδια η ενιαία αγορά. Θεωρώ ότι η προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι μηδαμινή. Και νομίζω ότι θα πρέπει μαζί να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Πρότεινα ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ίδιος, να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής και να δείξει ότι όντως η πολιτική αυτή της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των προτεραιοτήτων. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργείται και μια καλή διασύνδεση με το Συμβούλιο, όπου ανάλογη πρωτοβουλία θα αναλάμβανε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φτάσουμε ακόμα σε αυτό. Αν δείτε τι αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου, ουσιαστικά θα δείτε κάποιες πολύ σημαντικές προτάσεις. Από τη μια έχουμε την πράξη για την ενιαία αγορά του Επιτρόπου Μπαρνιέ και υπάρχουν και τρεις ακόμα προτάσεις οι οποίες αποτελούν τμήμα μιας γενικότερης στρατηγικής για την ενιαία αγορά για την οικονομική δηλαδή ολοκλήρωση. Έχουμε την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια της Επιτρόπου Ρέντινγκ, την επικοινωνία της Επιτρόπου Ντεγκούχτα του Επιτρόπου με για τις ανοιχτές αλλά όχι αφοπλισμένες αγορές και την έκθεση του κύριου Ταγιάννη, την πρωτοβουλία του κύριου Ταγιάννη για την βιομηχανική πολιτική. Βλέπετε ότι μέσω των προτάσεων αυτών προσπαθούμε να θεραπεύσουμε κάποια, έναν κατακαιρματισμό που είχαμε στην αρχή και προσπαθήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να κάνουμε μια πιο ολιστική, μια πιο σφαιρική πρόταση. Υπό το φως των πολύ σημαντικών προτάσεων που έκανε ο Επίτροπος Μπαρνιέ και προ όφελο των δικών σα προσπάθειών, πιστεύω ότι οι επόμενοι τέσσερι μήνε θα μπορούσαν να μα απασχολήσουν σε δύο επίπεδα. Πρώτον, αυτή η τετράμινη δημόσια διαβούλευση, η οποία σαφώ θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Θα είναι μια πολύ υγιής συζήτηση, το οποίο όμως δεν θα βοηθήσει σαφώς καθόλου τα προβλήματα τα οποία ήδη υπάρχουν και τα οποία πρέπει να ληφθούν με μια ταχύ ανάληψη νομοθετικών αποφάσεων. Πιστεύω επίση ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους τέσσερις αυτούς μήνες προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε κάποιους νέους πολιτικούς συμβασμούς. Είδαμε, κύριε Υπουργέ, ότι η Βελγική Προεδρία ήδη είναι πάρα πολύ ικανή και έκανε πολύ καλές σχετικές προτάσεις και ελπίζουμε ότι ακόμα και αύριο θα έχουμε ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Το έγγραφο του κύριου Μπαρνιέ δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο πώ θα καταφέρουμε να κάνουμε πιο αποδεκτή την ενιαία αγορά από τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως όσον αφορά τι κοινωνικές ανησυχίε που έχουν εκφραστεί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να τονίσουμε περισσότερο την ακόλουθη πτυχή, δηλαδή το συντονισμό των φορολογικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. παρουσιάζεται ως ένας τρόπος για να διευκολύνουμε καλύτερα την λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού είναι πολύ σημαντικό σαφώς, αλλά υπάρχουν και πολλοί πολίτες που πιστεύουν ότι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς χωρίς φορολογικό συντονισμό σιγά σιγά καταπνίγει την, τον ίδιο το ρόλο που διδραματίζει η απασχόληση εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός ο συναντισμός αυτός και θα πρέπει να τονιστεί ακόμα περισσότερο. Και χαιρετίζω το ότι στον τομέα αυτό, όπου οι περισσότεροι είπανε μην κάνετε απολύτως καμία πρόταση, δηλαδή να έχουμε μια ομάδα πολιτικής φορολογικής όπου θα απαρτίζεται από υπουργούς από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επικεφαλή στον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Φορολογία τα πράγματα εδώ πέρα κινήθηκαν πολύ θετικά. Έγινε η πρώτη τέτοια συνεδρίαση με επικεφαλή στον κύριο Σεμέτα και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθεί ακόμα περισσότερο αυτή η προσπάθεια. Αν λοιπόν έχουμε την πράξη για την ενιαία αγορά και τη συνδυάσουμε με το φορολογικό συντονισμό και εφόσον καταφέρουμε, προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενιαία αγορά με τα δύο αυτά μέσα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε και να επιλύσουμε τα προβλήματα και να τονίσουμε τα θετικά της ενιαίας αγοράς. Και θα καταφέρουμε επίσης να προωθήσουμε πολύ περισσότερο την εφαρμογή των νομοθετημάτων για την ενιαία αγορά. Έχουμε επίσης την πρόταση παριθμών 47 στην πράξη για την ενιαία αγορά για μια εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για να δημιουργηθεί μια πολιτική για την καλύτερη επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Εγώ στην εκθεσή μου έκανα κάποιες περαιτέρω προτάσεις όπως το να χρησιμοποιήσουμε κάποιους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης για την ε, μέγιστη διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάση, που όπως ε, γνωρίζετε προκαλούν πολλά προβλήματα στη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και επίσης ε, προτείνω να δούμε αν θα μπορούσαμε να ευθυγραμμίσουμε περισσότερα τα, συστήματα επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς με τα όσα απαιτούνται στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα. Να πούμε ότι η ανταγωνιστικότητα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κοινωνική ισότητα, γιατί ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα υποστηρίζει τους λιγότερο δυνατούς σε σχέση με τους πιο δυνατούς, σε σχέση με τις πλούσιε χώρε, σε σχέση με αυτού οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια μονοπωλίων. Επίσης συμφωνώ με αυτούς που πριν από λίγο είπαν ότι ε, θα μπορούσε να συμπληρώσει κατά αυτόν τον τρόπο πολύ καλά η πρόταση αυτή, την πράξη για την ενιαία αγορά. Αν δηλαδή μπορούσαμε να έχουμε στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς μια ευθυγραμμισμένη, συντονισμένη, ε, ένα συντονισμένο μέτρο για τις συλλογικές ε, προσφυγές. Ήμουν επίτροπος για την έννοια αγορά και συνέχεια επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού και όπως είναι σύνηθες για έναν επίτροπο αρμόδιο για την ενιαία αγορά, άρχισα να εργάζομαι για να προστατεύσω τους δημιουργούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταστρέψουμε την ε, ενιαία αγορά νομοθετώντας πάρα πολύ αυστηρά για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα συμφέροντα τα οποία έχουν παγιωθεί, συνεταιριστικά συμφέροντα, συντεχνιακά με συγχωρείτε συμφέροντα, και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια καλώς λειτουργούσα ηλεκτρονική ενιαία αγορά η οποία θα συμφιλιώσει τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους με τις αρχές της ενιαίας αγοράς και με την όλη ευρωπαϊκή οικοδόμηση η οποία δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται από ένα υπερβολικό σύστημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ καθηγητή Μόντι για την τολμηρή και πραγματιστική αντίληψη που έχετε για την εσωτερική αγορά, την ενιαία αγορά. Έχουμε λίγο χρόνο και πρέπει να είστε πολύ σύντομοι στις ερωτήσεις σας, γιατί σε λίγο θα πρέπει να ξεκινήσει το δεύτερο πάνελ. Λοιπόν, η κυρία Βερνιό, πρώτη ερώτηση. Θα είμαι πολύ σύντομη. Οι ερωτήσεις μου είχαν παραλείπει τον Επίτροπο Μπαρνιέ, αλλά λόγω της εμπειρογνωμοσύνης και της εμπειρίας την οποία συγκεντρώνει ο κύριος Μόντι και του το αναγνωρίζουμε αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορέσει να απαντήσει ελπίζω στην ερώτησή μου. Δεν θα επανέλθω στις υπηρεσίες καθολικού ενδιαφέροντος. Αλλά η πρόταση υπαριθμή 25 είναι ιδιαίτερα θα έλεγα αδιαυκρίνηστη και με ενοχλεί η διατύπωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την πρόταση υπαρήθμου 40, η πρόσβαση στις πιστοτικές τραπεζικές υπηρεσίες. Πολύ σημαντική πρόταση. Όταν ζητάμε να προσκαλέσουμε τον πιστοτικό τομέα να καταθέσει μια πρωτοβουλία αυτορύθμισης, Τώρα τι ακριβώς θέλετε. Μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια και τους προηγούμενους μήνες Πιστεύετε τώρα ότι μια τέτοια πρόταση επαρκεί έτσι ώστε να δώσει εμπιστοσύνη ο πολίτης στο τραπεζικό του σύστημα και να αποφύγουμε τις καταχρήσεις που γνωρίσαμε όλοι τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ κύριε Φερνιό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πάρω το λόγο θέτοντας μία ερώτηση στον κύριο Μπαρνιέ, αλλά μιας και δεν είναι εδώ θα τη θέσω στον κύριο Μόντι. Uh, αφορά το θέμα της συνεργασίας και του συντονισμού στον φορολογικό τομέα. Είπατε ότι εδώ υπάρχει χώρος για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά. Είναι κάτι το οποίο ε, ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες, είπατε, των πολιτών. Εδώ διαφωνώ μαζί σας. Το θέμα του συντονισμού στον συγκεκριμένο τομέα είναι ένα θέμα το οποίο ανακοινεί ανησυχίες πάρα πολλές στους πολίτες σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό επιβολής για τις επιχειρήσεις, ναι. Αυτό μπορεί να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο. Αλλά πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει ανάγκη εναρμονισμένου επίπεδου επιβολής ΦΠΑ σαν παράδειγμα σε όλες τις χώρες. Πιστεύετε ότι ο φορολογικός αυτός συντονισμός θα παίξει σημαντικό ρόλο στην παρούσα φάση, εφόσον θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει ανάγκη για ουσιαστική βελτίωση της εσωτερικής αγοράς. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μόντι, θα ήθελα εγκάρδια να σας ευχαριστήσω γιατί παρουσιάσατε μια σφαιρική αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει για τη λειτουργία της ε, εσωτερικής αγοράς και περνάω στη μητρική μου γλώσσα. Η εσωτερική αγορά ε, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα κατανοητό από τον πολίτη. Δεν κατανοεί ο καθημερινός πολίτης ποιο είναι το όφελος. Στα πλαίσια του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης ουσιαστικά βλέπουμε ότι ε, νιώθουμε υφιστάμεθα πιέσεις από πολλές πλευρές. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να έχουμε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και γι' αυτό είναι απαραίτητο όταν μιλάμε στον Ευρωπαίο πολίτη να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι για το τι μιλάμε. Αυτή η χρονική υστέρηση, η προθεσμία τεσσάρων μηνών για τη διαβούλευση είναι κάτι το απαραίτητο. Γιατί όχι. Παράλληλα με αυτό όμως Μου δημιουργείται η αίσθηση ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα στο μέλλον. Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι απόψεις των κρατών μελών για την, εσω... για την ενιαία αγορά. Υπάρχει, θέλουμε δεν θέλουμε, ένα σχετικό ποσοστό προστατευτισμού σε εθνικό επίπεδο. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το επίπεδο αυτό και τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν. Σύντομος ο επόμενος ομιλητής λέει ο πρόεδρος. Κύριε καθηγητά Μόντι, με εξέπληξε λίγο η διαφωνία σας σε ό,τι αφορά την μέθοδο που έχει επιλέξει η Κομισιόν υπέρ διαβούλευσης. Μπορεί να έχετε και δίκιο όμως. Ε, τα 50 μέτρα είναι γενικόλογα και δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε μαζί τους. Όλοι συμφωνούμε κατά βάση. Πολλοί δε περισσότερο που έχουν εν μέρει ήδη συζητηθεί. Αυτό που θα είναι δύσκολο είναι το επόμενο στάδιο. Γιατί αυτά τα μέτρα βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο εφαρμογής. Πρέπει να δούμε πού βρίσκονται για να καταλάβουμε πόσο γκάζι πρέπει να βάλουμε σε καθένα από αυτά τα μέτρα. Αλλά ακόμα πιο δύσκολη θα είναι η τρίτη φάση, το τρίτο θέμα, που θα είναι ο καθορισμός προτεραιοτήτων δράση. Έχουμε 50 μέτρα σε διαφορετικά επίπεδα, στάδια εφαρμογής, διαφορετικής δυσκολίας. Και χρειάζεται λοιπόν να καταρτήσουμε προτεραιότητες, να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε και τι θα μείνει για αργότερα. Εκεί θα προκύψουν πολλές διαφωνίες. Οπότε η δική μου ε, ε, πρόταση είναι η δική σας πρόταση, είναι και δική σας πρόταση, δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μόντι, καθηγητά Μόντι. Για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω την τιμή να δώσω απάντηση αντικαθιστώντας αυτόν που με διαδέχτηκε, <laughs> τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Κυρία Βερνιό, ε, δεν μπορώ να γνωρίζω τις σκέψεις του Μισελ Μπαρνιέ, παρόλο ότι οι γνώμες μας ε, συμπίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, πρόταση 40 αναφέρει η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση σε ορισμένες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες στην αρχή του 2011. Προφανώς συμφωνώ. Έτσι κι αλλιώς το είχα και εγώ προτείνει στην έκθεσή μου. Και στους έξι μήνες που έχουμε μεσολαβήσει δεν έχω αλλάξει γνώμη. Αλλά για να συστιαστούμε στο δεύτερο τμήμα κυρίω, λέει, θα υποβάλει τον ε, τραπεζικό τομέα σε μια πρωτοβουλία αυτορύθμισης για την ε, συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των ε, τραπεζικών επιβαρύνσεων. Οπότε εσείς αμφιβάλλετε για το κατά πόσο ο τραπεζικός τομέας θέλει ή πρόκειται να πράξει κάτι τέτοιο ο Μισελ Μπαχνιέ γνωρίζουμε πως ε, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος για το θέμα της, ε, των τραπεζικών ρυθμίσεων συνεπώς ε, για να το έβαλε εδώ θα έχει τους λόγους του να υπογραμμίσω επίσης και αυτή είναι δική μου προσωπική γνώμη ότι ασφαλώς και θα πρέπει να διορθώσουμε τις ε, σημαντικές αδυναμίες ρύθμισης του χρηματοοικονομικού τομέα που υπήρχαν από το παρελθόν αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, εκπαιδεύσουμε ή να επανεκπαιδεύσουμε τις ε, χρηματοοικονομικές αγορές να λειτουργούν ως αγορές. Συνεπώς δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή καμιά άλλη χώρα μπορεί να προχωρήσει ε, προγραμματίζοντας τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Συνεπώς η πρωτοβουλία της αυτορύθμισης είναι καλή. Αν μάλιστα αυτή την πρωτοβουλία την αναλάβει η Κομισιόν που έχει και νομοθετικές εξουσίες, προφανώς ο ενδιαφερόμενος θα την προσέξει. Τώρα για το συντονισμό των φορολογικών πολιτικών. Η ανησυχία είναι μήπως τελικά αυτό δεν ευνοήσει την εσωτερική αγορά. <laughs> Αλλά μετά είδα στην ομιλία σας ότι είσαστε πολύ πιο φιλόδοξος από μένα και από τον κύριο Μπαρνιέ. Γιατί λέτε, ίσως πράγματι υπάρχει, για, υπάρχει ανάγκη για ένα ελάχιστο φορολογικό συντελεστή των κερδών των επιχειρήσεων. <laughs> Αυτό είναι ένας πάρα πολύ φιλόδοξο στόχο για το σημερινό στάδιο τη Ευρωπαϊκή οικοδόμησης και τα περισσότερα κράτη-μέλη θα διαφωνούσαν. Ούτε εγώ δεν τόλμησα καν, αντίθετα με εσά, που έχω την εντύπωση ότι αντιτίθεστε με, την, ε, με το φορολογικό συντονισμό, ούτε εγώ δεν τόλμησα καν να προτείνω ένα τέτοιο φιλόδοξο ε, μέτρο. Μετά βέβαια για τον ε, ΦΠΑ λέτε ότι ίσως η λειτουργία της ιδιωτικής αγοράς χρειάζεται μια μεγαλύτερη ομοιομορφία της συντελεστών. Μετά, ε, η συνάδελφό σας ε, έθεσε το θέμα της ε, λειτουργίας πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα. Σίγουρα είναι σημαντική η συμμετοχή του κοινού, αλλά θα πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα να συνεργαστούν επίσης και τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν όλα, οπότε τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει το, έτσι ώστε να συμπέσουν αυτές οι απόψεις και να συγκλίνουν. Και ο καθηγητής Κορέα είπε ωραίο να έχουμε 50 προτάσεις αλλά θα πρέπει να καθορίσουμε και προτεραιότητες και να συμφωνήσουμε επί αυτών. Τι θα έκανα εγώ και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα οικοδομούσα πάνω στις διαβουλεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα. Για παράδειγμα, εγώ για κάθε κράτος μέλος έχω έναν πίνακα για το ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι κατά κάθε μιας από αυτέ τι προτάσει που επέβαλα εγώ και που συμπίπτουν κατά βάση σε μεγάλο βαθμό με τι προτάσει του κ. Μπαρνιέ. Έχω του αντίστοιχου πίνακε για όλε τι πολιτικέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι υπέρ, ποια είναι κατά. Υπάρχουν και κάποιες βέβαια ε, εθνικές απόψεις και παραλλαγές μέσα σε κάθε πολιτική ομάδα. Τα έχω λάβει όλα αυτά υπόψη και τα έχω καταγράψει. Συνεπώς έχει ήδη γίνει μια μεγάλη δουλειά διαβούλευσης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Συνεπώς, έχουμε ένα ημιτελές προϊόν ως αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε πάνω σε αυτό περαιτέρω συγκλήσεις. Ευχαριστώ τον καθηγητή Μόντι. Οι φιλελεύθεροι έχουν ζητήσει το λόγο. Νομίζω ότι για να κρατήσουμε τις ισορροπίες θα δώσουμε το λόγο στον κύριο για να θέσει μια συμπληρωματική ερώτηση σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μόντι. Πολύ συγκεκριμένε είναι οι απαντήσει τι οποίες ε, δώσατε σχετικά με την τετράμινη περίοδο. Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι η προθεσμία αυτή δεν είναι αρκετά φιλόδοξη δεν θα μας καλύψει πλήρως και ε, νομίζω ότι ε, και τα μέσα ενημέρωση δεν ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα και αυτό μας εκπλήσει γιατί έχουμε δαπανίσει πολλή ενέργεια γύρω από αυτό και είναι περίεργο το να βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος που να ενδιαφέρεται. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποια άλλα στοιχεία Αναφέρθηκε το θέμα της Burning Platform. Θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα το συγκεκριμένη, το, τη συγκεκριμένη αυτή πλατφόρμα έτσι ώστε να έχουμε κάτι να προτείνουμε. Θα ήθελα κύριε Μόντι να μου διευκρινίσετε λίγο τις απόψεις σας γύρω από αυτό. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα και στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ίσως να μπορέσουμε να παίξουμε έναν βασικό ρόλο για να πιέσουμε και τα άλλα επίπεδα λήψη αποφάσεων. Κύριε Μόντι, συμπληρώστε. Um, by the way, Mr. Chairman, uh, Δεν είδα ότι είχατε επιστρέψει κύριε Χάρμπορ, γι' αυτό δεν σας ανέφερα στο χαιρετισμό μου. Πράγματι αυτή η πρωτοβουλία οφείλει πολλά σε εσά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, συμπληρώνει ο κύριος Μόντι, ότι ε, λέμε τα ίδια πράγματα. Λέει προς τον κύριο Λόκεργκάρτ. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινοβουλευτική σας επιτροπή. Έχετε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προτάσεις και με αρκετή επιτυχία και έχετε τονώσει την πολιτική ορατότητα ενός θέματος το οποίο θα έλεγα δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που του πρέπει. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα ικανοποιήσει μόνο αυτούς οι οποίοι προωθούν συγκεκριμένα θέματα. Αλλά εάν τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η κοινή γνώμη δεν θεωρεί ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, τότε η πρωτοβουλία αυτή είναι φυσιολογικό ότι δεν θα προχωρήσει. Ελπίζω λοιπόν και το είπα και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος με τίμησε ζητώντας μου να προετοιμάσω την έκθεση αυτή υποσχέθηκα ότι θα είμαι απόλυτα ευθύς και ειλικρινής και του είπα και προφορικά ότι θα υπάρξει τεράστια προστιθέμενη αξία αν ο ίδιος σαν πρόεδρος της Επιτροπής αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία. δεν ανήκει στην πολιτική. Δεν θα έλεγα, δεν είναι η ναυαρχίδα αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρώπη του 2020 γιατί δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μία σημαία, χρειάζεται πολλές. Λοιπόν δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα να προκαλέσω τη συνάδελφό μου την κυρία Τού να προεδρεύσει της επόμενης συνάντησης, του να προεδρευσει τη επόμενη συνάντηση του επομενου πανελ Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε Γκρέχ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριε Μόντι, είναι μεγάλη τιμή να σας καλωσορίσουμε σε αυτήν τη συνάντηση για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και τους δύο ομιλητές τον κύριο Λιβιέ Σαστέλ και τον κύριο Φάμπιον Τσούσλι. Ήδη τους παρουσίασε τον κύριο Σαστέλ και τον κύριο Τσούλιγκ ο Μάλκομ Χάρμπορ. Η ιδέα της οργάνωσης αυτού του φόρουμ που είχα προτείνει στα πλαίσια της συζήτησης ε, για τον ε, Ευρωπαϊκό Πίνακα Βαθμολογίας έτυχε θετική υποδοχή και από του συναδέλφου μου στο Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Μπαρνιέ για την προσωπική του συμμετοχή και αφοσίωση. Όπως λέει και η πρόταση 44 της ενιαίας πράξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τακτικά θα εξετάζει την κατάσταση της ε, ενιαίας αγοράς σε συνεργασία με τους υπολείπους εταίρους οργανώνοντας κάθε χρόνο ένα φόρουμ για την ενιαία αγορά μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους εκπροσώπους των υπολείπων οργάνων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όλους τους άλλους εμπλεκομένους. Κύριε Μόντι, θέσατε την εσωτερική αγορά στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πολίτης πρέπει να ενδιαφερθεί και θα τον οδηγήσουμε σε αυτό, θα τον βοηθήσουμε σε αυτό. Κάνουμε μια προπαρασκευαστική δουλειά που θα είναι ελπίζω αποτελεσματική. Βλέπουμε και άλλες προτάσεις στην ενία πράξη. Σωστή στενή σχέση με τα κράτη-μέλη, διαβουλεύσεις με την λεγόμενη κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, για τη σωστή ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων των κανόνων για τους κανόνες της νέας αγοράς. Η παρουσία εδώ του Υφυπουργού Κόρολετς δείχνει πόσο και η επερχόμενη Πολωνική Προεδρία ενδιαφέρεται για το θέμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω επίσης και τους πάρα πολλούς φιλοξενούμενους από διάφορες οργανώσεις της Κρακοβίας όπου θα γίνει το επόμενο φόρουμ από τη Βαρσοβία, από το Μάστριχτ και από πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Όλοι αυτοί οι νέοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης δείχνουν με την παρουσία τους την επιθυμία τους να πάρουν μέρος στη διαδικασία αυτή και να διαμορφώσουν την ενιαία αγορά είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τις δικές μας ευθύνες των μελών δηλαδή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους τους φίλους και συναδέλφους να χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να βοηθήσουμε το κοινό να συνειδητοποιήσει τα θέματα της ενιαίας αγοράς σε όλα τα κράτη-μέλη. Το επίπεδο της μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως επίσης και τα προγράμματα μεταφοράς κοινοτικής νομοθεσίας, που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συζητηθούν. Περαιτέρω τακτικές συναντήσεις των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανάμεσα στα κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι η πράξη της ενίας αγοράς σίγουρα θα βοηθήσει και την προώθηση της ίδιας τη ενία αγορά, η οποία δεν είναι μία βίβλος όπως είπε ο κ. Μπαρνιέ και σε κάποιου τομεί υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης. Θα πρέπει λοιπόν να διαβολευτούμε με τους πολίτες, ξεκινάμε τώρα αυτή τη διαβούλευση. Πρέπει να βελτιώσουμε την ενία αγορά. Απαιτείται να γίνει πιο αποδοτική. η στόχοι μας πρέπει να είναι πιο σωστοί. Είναι σημαντικό να μειώνουμε το έλλειμμα της μεταφοράς της νομοθεσίας στην εθνική, αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχουν και άλλα που πρέπει. Τα benchmarks, σαν παράδειγμα, για διαδικασίες επί παραβάση, που είναι διαδικασίες οι οποίες είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες. Κύριε Μόντι, έχετε δίκιο. Πρέπει να ταξινομήσουμε τις ευθύνες και να τακτοποιήσουμε τις ευθύνες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι συλλογική μας ευθύνη. Απαιτείται να γίνει μια συλλογική προσπάθεια έτσι ώστε η ενιαία αγορά να γίνει πιο λειτουργική για όλους, για όλους τους πολίτες, για όλους εμάς. Και αυτή η προσπάθεια την έχουμε αναλάβει εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα θα ήθελα πλέον να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Βελγικής Προεδρίας, τον κύριο Ολιβιέ Σαστέλ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι βουλευτές και αγαπητοί συνεργάτες, είναι μεγάλη τιμή για μένα που παίρνω το λόγο εδώ με την ευκαιρία του πρώτου φόρουμ για την ενιαία αγορά. Γνωρίζουμε όλοι μας και όλες μας τις προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τα επόμενα 10-20 χρόνια. Για να ανταποκριθούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 και γνωρίζουμε ότι η νέα αγορά είναι ένα πλεονέκτημα αλλά ταυτόχρονα και ένα απαραίτητο εργαλείο αυτής της στρατηγικής. Τόσο αυτή η στρατηγική όσο και η νέα αγορά δεν ε, θα πρέπει να περιορίζονται σε δηλώσει προθέσεων. Χρειάζονται συγκεκριμένες ε, δράσεις και σίγουρα, μόλι το είπαμε, μια καινούρια ενισχυμένη ε, ε, ε διαχείριση. η, η πανική της αγοράς χρειάζεται να απαιτεί από εμά να αναλάβουμε σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό, μια καινούργια δέσμευση. Όλοι μας χρειαζόμαστε στην προσπάθεια αυτή. Ε, μιλώ εκ μέρους του εξ του Πρόεδρου του Συμβουλίου και θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και κυρίω τον Πρόεδρο Μάλκον Χάρμπορ που ξεκίνησε αυτή την δημόσια συζήτηση για την νέα αγορά. Η ευθύνη που μας ε, βαρύνει είναι μεγάλη για να γεννηθεί ξανά ο διάλογος ε, και να συμμετέχουμε όλοι συλλογικά αποτελεσματικά στην εφαρμογή της ε, πράξης για την νέα αγορά στο τέλο του 2012. Η, τον ανακοίνωση 28 Οκτωβρίου 2010 που παρουσίασε ο Επίτροπος Μπαρνιέ στο προηγούμενο πάνελ ε, έχει στο τρίτο κεφάλαιο 7 προτάσεις εργαλείων από, τις, από την 44 έως την 50 για να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση ε, της ε, ε νέας αγοράς. Το Συμβούλιο, όπω γνωρίζετε, δεν έχει λάβει θέση επί αυτής της ανακοίνωση. Ε, Συνεπώ, αυτά που ακούτε από μένα είναι προκαταρκτικά και δεν δεσμεύουν τα κράτη-μέλη. στόχο μα είναι να υιοθετήσουμε συμπεράσματα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα στις 10 Δεκεμβρίου επί Βελική Προεδρία. Αυτά τα συμπεράσματα σίγουρα θα σχολιάζουν και τα εργαλεία που θα είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ε, εσωτερική αγορά. Πιο συγκεκριμένα όμως, ας δούμε μερικέ από αυτέ τι ε, προτάσεις με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενό καινούριου πλαισίου διαλόγου για την εφαρμογή των κειμένων αυτών προ όφελο των βασικών δικαιούχων που είναι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Ας ξεκινήσω με την πρώτη πρωτοβουλία καλή διακυβέρνηση που είναι η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση. Είναι παρθμό 44 πρόταση. Στην έκθεση του Ιανουαρίου 2010, η Κομισιόν ΙΜΚΟ του Κοινοβουλίου είχε προτείνει τη διοργάνωση ενό ετήσιου φόρουμ ενιαία ε, αγορά. Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να ξεκινήσει προκειμένου να προωθηθεί μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και μια πραγματική δέσμευση, προσήλωση ε, υπέρ τη μεταγραφή και τη εφαρμογή ε, τη ε, νομοθεσία σχετική με την εσωτερική αγορά. Η ύπαρξη ενό δραστήριου δικτύου που θα διαρθρώνεται σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικό, διοικητικό, κοινοβούλια, εταιρείε, κοινωνία των πολιτών θεωρείται ω στρατηγική σημασία προκειμένου να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Μετά, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εκτελεί μια αμοιβαία αξιολόγηση μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή και ε, μεταγραφή της οδηγίας υπηρεσιών. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει και μια δημόσια διαβούλευση των stakeholders, των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται από αυτήν την οδηγία μεταξύ του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 2010. Η, τα αποτελέσματα αυτής της ε, ε, διαδικασίας διαβούλευσης θα περιληφθούν σε μια έκθεση Κομισιόν που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν το τέλος του 2010. Υποθέτω ότι θα ξεκινήσουν συζητήσεις για αυτό το θέμα από το 2011 και μετά προκειμένου να ανταλλάξουμε τις καλές πρακτικές και να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Καλό είναι επίσης να υπενθυμίσουμε τη σημασία της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών για το μέλλον της ίδιας της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Μετά, πρώτα 45 διεύρυνση του συστήματος ε, πληροφοριών της εσωτερικής ε, αγοράς, το IMI. Πίσω από αυτά τα αρχικά, το αρκτικό λεξο, βλέπουμε ένα σύστημα πληροφοριών τη εσωτερική αγορά. Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πολύγλωσσο που έχει ως στόχο να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών ε, και τη συνεργασία ανάμεσα στι διοικητικέ αρχέ των χωρών μα. Το IMI συνδέει τις διοικητικές υπηρεσίες και ενισχύει το διάλογο επιτρέποντας την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών ε, και την συνδρομή, αμοιβαία συνδρομή στο εσωτερικό της εσωτερικής αγοράς. Ε, δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη για να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα. Η επιτυχία της πρώτης ε, δοκιμαστικής φάσης του IMI στην ε, στο σύστημα ηλεκτρονικής υγείας της, ε, ε, και στα επαγγελματικά προσόντα μας οδηγεί στο να το διευρύνουμε και να το εφαρμόσουμε σε άλλους τομείς. Νομίζω ότι αυτό θα το δεχτεί θετικά το Συμβούλιο. Πρόταση 47 έχει ως ε, στόχο ένα μέγιστο 0,5% ελλείμματος στην μεταγραφή των νομοθετικών κειμένων ε, και που έχει σχέση με τον πίνακα αποτελεσμάτων, το βαθμολόγιο. Ε, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταγράφουν ορθά και μέσα στις προθεσμίες της, οδηγίας, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ε, ανεξαρτήτως παρόλων, παρόλων μάλιστα, παρόλες τις διαφορές στο μέγεθο την οργάνωση και την δομή των κρατών μελών ε, ανάλογες λύσεις ε, αλλά με τρόπο πιο ευέλικτο θα πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προβλήματα μεταγραφής. Το πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς και η κατάσταση κριτηρίων που θα περιορίζουν την, το έλλειμμα της μεταγραφής θα δράσουν θετικά σε αυτή τη διαδικασία μεταγραφής. Ο 21ος ε, πίνακας αποτελεσμάτων εταιρική αγορά που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο 2010 ε, αναφέρει ένα μέσο όρο 0,9% καθυστέρησης ή ε, ελλείψεων στην μεταγραφή των ευρωπαϊκών οδηγιών εταιρικής αγοράς. Αυτό αποτελεί σημαντική επιτυχία γιατί ε, έτσι σεβόμαστε την, τον κανόνα του μέγιστο 1%. Παρ' όλα αυτά ο μέσος όρος καθυστέρησης ε, μεταγραφής των οδηγιών είναι ψηλός και υπάρχει και το θέμα της ε, συμφωνίας μεταξύ των εθνικών κειμένων Πάντω ε, σε ένα ιδανικό κόσμο ε, θα έπρεπε να μειωθούν οι ε, καθυστερήσει και ενδεχομένω το 0,5% ενδεχομένως όμως το 0,5% θα είναι δύσκολο να το σεβαστούμε. Το να απαιτούμε πίνακες αποτελεσμάτων για κάθε οδηγία ε, δεν βρίσκει σύμφωνο όλο το Συμβούλιο, το γνωρίζετε αυτό. Γι' αυτό αυτή η πρόταση δημιουργεί φόβους ότι θα καθυστερήσει η μεταγραφή, ότι θα γίνει πιο περίπλοκη η εφαρμογή των οδηγιών από τα ομόσπονδα κράτη και ότι θα είναι και πιο επαχθής ε, οικονομικά. Ως προστάτη των ε, θεματοφύλακας των συνθήκων η Κομισιόν έχει την πρόθεση να προχωρήσει πιο γρήγορα ε, και να ζητήσει τα κράτη-μέλη να σέβονται πιο πολύ τις ε, προθεσμίες ε, μάλιστα ε, όμως ε, ένας αριθμός αποφάσεων δημιουργεί το κίνδυνο να αυξηθούν οι καθυστερήσεις. Η Προεδρία του Βελγική Προεδρία οργανώνει 22-23 Νοεμβρίου μια, ένα συνέδριο για την μεταγραφή των ευρωπαϊκών οδηγιών. Έχει ως στόχο να ανταλλαγούν οι καλές πρακτικές και να προτείνει συμπεράσματα τα οποία θα επέτρεπαν στα κράτη-μέλη να βελτιστοποιήσουν τα συστήματα μεταγραφής των ευρωπαϊκών οδηγιών. Σε ό,τι αφορά τις ε, διαδικασίες επί παραβάση, ε, γνωρίζουμε, ιδιαίτερα εμεί στο Βέλγιο, ε, ότι είμαστε στον πάτο ουραγίτ στην καταταξή διότι έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πάντω ε, είναι καλό να υπογραμμίσουμε ότι για ορισμένε διαδικασίε επί παραβάση οι παρατηρήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν αμφισβητηθεί στη, από νομικής πλευράς από τα κράτη-μέλη. Ενώ σε άλλε περιπτώσει τα κράτη-μέλη περιμένουν την αντίδραση κομισιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα ε, και παρόλα αυτά, όλες αυτές, παρόλο ότι περιμένουν την Κομισιόν, ε, οι περιπτώσεις αυτές καταγράφονται και προστίθενται στο αποτέλεσμα. Ε, γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και άτυπα ε, εργαλεία όπως το EU Pilot και το Solvit. Τέλος θα ολοκληρώσω αυτό το κεφάλαιο λέγοντας ότι το βαθμονόμιο της εσωτερικής αγοράς δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα μέσο πίεσης, θα πρέπει να χρησιμεύει και στο σύστημα πληροφόρησης και στο, στην πρόθεση του διαλόγου με τα κράτη-μέλη. Το, η πρόταση 49 λέει ότι θα πρέπει ε, να επικοινωνούμε καλύτερα και να προωθήσουμε την ενιαία θηρίδα και το, το πόρταλ «Η Ευρώπη σας ανήκει». Ο, ο Ζων Ρέι το έλεγε η, «Η Ευρώπη παραπονιέται και το ξέρει, η Ευρώπη πραγματοποιείται και το ξεχνάει, το αγνόει». Ε, από 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν σε μια χώρα, ευρωπαϊκή χώρα που δεν είναι η δικιά τους και αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ε, Διαπιστώνουμε όμως ότι δεν είναι ενήμεροι, πλήρως ενήμεροι για τα δικαιώματα αυτά ή αντιθέτως είναι ε, παραπληροφορημένοι και νομίζουν ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα από όσα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι αποτελεσματικά ενημερωμένοι για το τι μπορεί να κάνει ή δεν μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, εργαλεία ε, βοήθεια, συνδρομη ε, ενημέρωση υπάρχουν και λειτουργούν. Διαπιστώνουμε όμως σήμερα ότι ακόμα και οι γνώστες, οι μοιημένοι, δύσκολα βρίσκουν το δρόμο τους ε, σε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε λαβύρινθο των δικτύων πληροφόρησης, συνδρομής, γενικευμένων ή πιο ειδικευμένων ή ακόμα και στα site πληροφόρησης εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν θέλει να τα ομαδοποιήσει, να ομαδοποιήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε ένα κοινό πόρταλ ε, ε, του οποίου το, το ε, interface θα είναι η σελίδα Ευρώπη σας ανήκει. Ε, ε, είμαι πεπισμένος ότι θα συνειδητοποιήσουμε καλύτερα το, την ουσιαστική αγορά αν βελτιώσουμε την πληροφορία και την ε, συνδρομή και με άτυπους τρόπου όταν αυτό χρειάζεται. Ο λόγο είναι πολύ απλός. Ε, όλοι μας, μας, μας, μας ενδιαφέρει η Ευρώπη να κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιώσει, για παράδειγμα, να διευκολύνει την κινητικότητά μας, ε, τακτική ή μη, δεν έχει σημασία, θα είμαστε σε θέση να προσωριζόμαστε τα δικαιώματά μας όταν έχουμε ήδη εργαλεία και έχουμε, απλά πρέπει να γίνουν πιο προσβάσιμα στο ευρύ Η Βελική Προεδρία ε, συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία βάζοντα ε, στο, ε, επίσημο site της Προεδρίας για έξι μήνες Συγκεκριμένε πληροφορίε, εύχριστε για τις πηγέ πληροφοριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τις επιχειρήσεις και του ευρωπαίους πολίτες. Πρωτοβουλίες όπω το καινούριο πόρταλ «Η Ευρώπη σα ανήκει» που δει πληροφορίε ανάλογα το προφίλ του χρήστη ε, έχουν σημαντικό δυναμικό. Επίση, δίκτυα όπω το Solvit ή το Ευρωπαϊκό ε, Κέντρο Καταναλωτών ε, βοηθούν έτσι ώστε να προσανατολίζεται ο χρήστη στον κατάλληλο συνομιλητή. Η, η Βελική Προεδρία πιστεύει ότι είναι χρήσιμο ε, να ενισχύσουμε την γνώση αυτών των εργαλείων έτσι ώστε ε, να απομυθοποιηθεί η ευρωπαϊκή δράση. Πρόταση 50 έχει ως ε, στόχο να εδρεωθεί το Project EU Pilot και να ενισχυθεί το δίκτυο Solvit. Το EU Pilot δίνει την ευκαιρία να λύσουμε τα προβλήματα της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης άτυπα και να αποφύγουμε ε, διαδικασίες επί παραβάση. Ε, αυτή τη στιγμή τρία κρατημέλη είναι εκτός ε, του EU Pilot, μεταξύ αυτών το Βέλγιο, οι οι αρχές μας θα αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουμε από την 1η Πρώτη του 2011. Ε, υπάρχει και το δίκτυο Solvit, γνωρίζετε είναι μια υπηρεσία ε, που ε, λύνει πολλές φορές διαμεθοριακά προβλήματα των πολιτών μας στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής αγοράς. Το τρίτο πάνελ θα δώσει την ευκαιρία να εξοικειωθούμε με αυτά τα εργαλεία, με την με το συντονισμό του Κριστιαν Μπουζόη που ε, ε, ήταν ο συντάκτης της ε, πρώτης πρότασης, μη νομοθετικής πρότασης για το Solvit. Το Solvit είναι ένα πολύ επιτυχημένο εργαλείο επίλυσης, μη εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών. Δεν, έχει, έχει, έχει μεγάλο δυναμικό, είναι επιτυχημένο στην αρχή του, πρέπει να ενισχυθεί και έχει βοηθήσει ήδη να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους διάφορους εταίρους και χρήστες. Η Βελική Προεδρία λοιπόν δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρόθεση αυτού του εργαλείου και χαίρεται που το επόμενο workshop Solvit θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 24 και 25 Νοεμβρίου αυτού του χρόνου ε, στο πλαίσιο της εβδομάδας ε, που θα αφιερώνεται στην μεταγραφή και την εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, κύριε και κύριοι, κύριε Υπουργέ, Κυρίε και κύριοι, ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του 2012 θα μπορούμε όλοι μας να λέμε ότι η ενιαία αγορά έχει πραγματοποιηθεί χάρη στη δική σας συμμετοχή, χάρη στη δική σας στήριξη. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαστέλ. Ο κύριος Φαμπιαντσούλα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά. Μια πολύ καλή πρωτοβουλία κατά την άποψή μου. Θα σας μιλήσω για το μέλλον. Ουσιαστικά το ερώτημα που θέτω είναι η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς αντιστοιχεί στην μελλοντική οικονομία της γνώσης και θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Να σας πω καταρχάς ότι η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων καθώς επίσης και η βελτίωση της διακυβέρνησης προτείνουμε είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για να πετύχουμε μια νέα ψηφιακή εσωτερική αγορά και πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό, σημαντική βάση για τις μελλοντικέ εξελίξεις. Τα όσα προτάθηκαν λοιπόν μέχρι στιγμής πιστεύουμε ότι ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν σε μια πιο ισχυρή εσωτερική αγορά, ιδίω για τις υπηρεσίες και στις οποίες θα μπορούσε να βασιστεί και η μελλοντική ψηφιακή ενία αγορά. Στο European Policy Center έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα της ψηφιακής ε, ενίας αγοράς και θεωρούμε ότι η ψηφιακή ενία αγορά μπορεί να επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα για όλη την Ευρώπη. Δεν θα αποφεληθούν μόνο οι επιχειρήσεις, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και μπορεί να βοηθήσει όμως και το κοινό, τους πολίτες. για ποιο λόγο πρέπει τα πράγματα να εξελιχθούν, μα γιατί αλλάζει η ίδια η οικονομία της Ευρώπης. Αν δούμε τον κόσμο γύρω μας, βλέπουμε ότι η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο μας πάρα πολύ γρήγορα. Η τεχνολογία διέπει πλέον όλους τους τομείς της κοινωνίας και όλους τους τομείς της οικονομίας. Βλέπουμε νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες στον ψηφιακό αυτό νέο κόσμο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και νέα φαινόμενα, όπως ο ψηφιακός αποκλεισμός. Η παγκοσμιοποίηση συνεχίζει και επηρεάζει βέβαια την οικονομία της Ευρώπης. Έχουμε όλο και περισσότερες παγκόσμιες αλυσίδες αξιών, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως στην ε, εικονική πλέον οικονομία, την ψηφιακή. Η γνώση και οι δεξιώσεις αποτελούν ε, ένα σημαντικό ταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και μας απασχολεί ακόμα περισσότερο το ζήτημα της εξωτερικής ανάθεσης της υπεργολαβίας που παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη. Επίσης, Υπάρχουν και νέοι τρόποι εργασία πλέον, εργασία από το σπίτι, συμβάσει που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα project, αυτοαπασχόληση και αλλάζουν σιγά σιγά τα όρια ανάμεσα στον δεύτερο χρόνο και την εργασία. Αλλάζουν όμω και επιχειρήσει. Βλέπουμε νέα επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία αναπτύσσονται. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται όλο και περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό θα συνεχιστεί άλλωστε. Και βλέπουμε ότι η γνώση αποτελεί πλέον πλεονέκτημα και περιουσιακό στοιχείο, θα λέγαμε, για όλες τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά του συνόλου της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία μετατρέπεται, αλλάζει και θα επιφέρει και νέες επιπτώσεις. Θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν και η νέα αγορά για να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις. Αν δεν τροποποιήσουμε τα πράγματα, τότε οι κανόνες της νέας αγοράς δεν θα είναι πλέον ρεαλιστικοί. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση της νέας αγοράς, η οποία να συνάδει με την οικονομία της γνώσης. Κατά την άποψή μα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει απλώ παθητικά να εξαλείφουμε τα εμπόδια, αλλά θα πρέπει να οικοδομήσουμε ενεργά την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να έχουμε κάποια θετικά μέτρα και μια καλύτερη εναρμόνιση, κυρίω για του πολίτε και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σταθερό συνεκτικό περιβάλλον. Διαφορετικά δεν έχουν καμία διάθεση να συμμετέχουν. Δεν θα πρέπει να έχουμε απλώ μια ελεύθερη μετακίνηση των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών και κατ' επέκταση και μια ελεύθερη μετα... κυκλοφορία της γνώσης. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η γνώση. Αποτελεί παράγοντα παραγωγής, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και η γνώση μεταδίδεται μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων βέβαια, εν υπάρχει στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο και με την ηλεκτρονική οικονομία, ηλεκτρονικές τραπεζικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επίση, το ανθρώπινο κεφάλαιο γίνεται όλο και πιο κρίσιμο. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τι δυνατότητε μετακίνηση και κυκλοφορία των εργαζομένων. Όταν μιλάμε για κυκλοφορία, μετακίνηση υπηρεσιών, αφαιρόμαστε και στην ελεύθερη κυκλοφορία βέβαια των ατόμων. Έχουμε κάποιε νέε προκλήσει και κάποιε προκλήσει που έχουν ανανεωθεί. Υπάρχουν κάποιοι τα δύσκολοι από πολιτικής πλευράς χώροι τους οποίους θα πρέπει να, με του οποίου θα πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με το ψηφιακό έγκλημα, τι γίνεται στο διαδίκτυο για το οποίο δεν υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ένας μεγάλος κατακαιρματισμός ακόμα στον τομέα αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν οι κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη, να ρυθμίσουν και να φορολογήσουν αποτελεσματικά τις ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο μόνο σε εθνικό επίπεδο. Πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού ψηφιακού τομέα. Πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε επιχειρήσεις κλίμακος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Το έχουμε πετύχει αυτό. Στον τομέα όμως της νέας οικονομία υστερούμε, για παράδειγμα στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Η ψηφιακή ενιαία κατά την άποψή μας αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή παραγωγικότητα και κοινοτομία και μπορεί να προσθέσει ένα 4% στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ μέχρι το 2020 αλλά ενδεχομένω να καταφέρει να συμβάλλει και ακόμα περισσότερο. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι η ψηφιακή αυτή οικονομία είναι ένα παράγοντα που θα συμβάλλει και στην έξοδο από την κρίση. Δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα μόνο στην καινοτομία και την παραγωγή στον τομέα της πληροφορικής, αναφερόμαστε σε όλους τους τομείς της οικονομίας που θα μπορέσει μέσω της τεχνολογίας να βελτιωθεί. Υπάρχουν και πολλά άλλα θετικά μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως η δημογραφική πρόκληση, ή κλιματικές αλλαγές. Όλο και περισσότερο έχουμε πολίτες οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες ε, προσδοκίες και που περιμένουν να αναπτύξουμε εμείς περισσότερο την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ιδίω οι νέοι έχουν τέτοιες απαιτήσεις. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι νέοι για ποιο λόγο δεν γίνεται διασυνοριακά να αγοραστούν ορισμένα προϊόντα, για ποιο λόγο δεν μπορούν να κατεβάσουν απόλυτα ελεύθερα τη μουσική ή τα έργα τα οποία θέλουν. Επίση, υπάρχουν πολλοί πολίτε που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλεια και προστασία στο ίντερνετ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ανταποκριθεί σε όλε αυτέ τι απαιτήσει και ανησυχίε. Ποιε είναι οι συστάσει μα τώρα, Δεν μπορώ να τι καλύψω όλε, δεν έχουν απαραίτητο χρόνο. Πολλά από αυτά τα οποία πιστεύουμε και εμεί έχουν καλυφθεί από τη σημερινή συζήτηση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί πολιτική έμφαση στην ενιαία αγορά και στην ψηφική ενιαία αγορά ιδιαίτερω. Πέρα από την έκθεση Μόντι και πέρα από αυτά που είπε ο καθηγητή Μόντι, ελπίζουμε ότι ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει τι νέε αυτέ πρωτοβουλίε. Χρειάζεται η απαραίτητη ηγετική θέση πυγμή προκειμένου να προωθήσουμε τι νέε αυτέ προτάσει. Το ζήτημα τη εμπιστοσύνη επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εμπιστοσύνη που θα δείχνουν οι πολίτε. Θέλουμε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο να συνάδει με την ε, οικονομία της γνώσης. Πρέπει επίσης να θέσουμε την απαραίτητη δομή, να δημιουργήσουμε την απαραίτητη υποδομή για την ε, νέα τεχνολογία της γνώσης. Αναφέρομαι για παράδειγμα στις εμπριζονικές υπηρεσίες. Όλες αυτές τις προτάσεις μπορείτε να τις δείτε στη δημοσίευση που έχουμε κάνει και θα σας δώσω και την ηλεκτρονική διεύθυνση στο τέλος της παρουσίασής μου. Είχαμε σαφώς κάποια σημαντική ηγεσία η ενιαία αγορά νίκη στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μπαρόσο το έχει πει αυτό πολλές φορές. Είχαμε βέβαια, έχουμε και την καταπληκτική έκθεση Μόντι και θεωρούμε ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας ότι μας δόθηκε δυνατότητα να συμβάλλουμε στην σύνταξη της έκθεσης αυτής. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν ε, πολλέ σημαντικέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προωθούνται αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλε προτάσει όπω αυτή για την βιομηχανική πολιτική. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέσα σε όλε αυτέ τι προτάσει υπάρχει ένα κίνδυνο κατακαιρματισμού αν δεν επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο συντονισμού. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι θα ληφθεί απαραίτητη δράση ταυτόχρονα σε όλου αυτού του τομεί. Δεν αρκεί να προωθούμε, να έχουμε πρόοδο σε έναν μόνο τομέα. Αν πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή ενιαία αγορά, πρέπει να σημειώνουμε πρόοδο ταυτόχρονα σε πάρα πολλού τομεί και η πρόοδο αυτή θα πρέπει να επέλθει πολύ γρήγορα. Ήδη υστερούμε σε πολλού τομεί Ακόμα όμω υπάρχει μπροστά μα η δυνατότητα να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά αυτή η δυνατότητα όλο και μειώνεται. Η υφιστάμενη πρόταση αναφέρεται σε πάρα πολλού τομεί, σε πάρα πολλέ πτυχέ. Παρ' αυτά χρειαζόμαστε περισσότερε λεπτομέρειε. Λέγεται σε πάρα πολλά σημεία τη έκθεση ότι πρέπει να επιτευχθεί στον ένα ή τον άλλον τομέα πρόοδο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε πώ ακριβώ θα επιτευχθεί αυτή η πρόοδο. Χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένε λοιπόν προτάσει και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε την περίοδο τη διαβούλευση για να κάνουμε ορισμένε προτάσει λίγο πιο συγκεκριμένε, λίγο πιο απτέ. Υπάρχει τώρα αρκή, ολοκλήρωση σε όλες τις ε, σε όλου του τομεί πολιτική. Αυτό μόνο ο χρόνο θα το αποδείξει. Το σημαντικό είναι υπάρχει όμως ένα κοινό όραμα, κάτι το οποίο θα φέρει μαζί τι διαφορετικέ διευθύνσει Ευρωπαϊκής Επιτροπή, του διαφορετικού ενδιαφερομένους, κάτι το οποίο θα συγκεράσει τις προσπάθειες. Δεν ξέρω βέβαια αν ε, ο βαθμός ε, φιλοδοξίας είναι αρκετά ισχυρός. για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που ακούστηκε πριν από λίγο. Αυτό το οποίο έχει σημασία εν τέλει δεν είναι τόσο οι προτάσεις όσο το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, στο γης μέλλον θα έλεγα, όλοι οι παράγοντες της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να θεωρούν ότι ανήκουν σε μία ενιαία κοινή αγορά και ότι δεν κινούνται σε μια κατακαιρματισμένη εθνική τελικά αγορά όπου υπάρχουν πάρα πολλοί φραγμοί και πάρα πολλές τάσεις προστατευτισμού. Αν δημιουργηθεί αυτή η πραγματικά ενιαία αγορά χωρίς εμπόδια, τότε τόσο στον πραγματικό όσο και στον εικονικό κόσμο θα είμαστε σε θέση πραγματικά να αποτιμήσουμε την μελλοντική επιτυχία της πράξης για την ενιαία αγορά και των υπολείπων προτάσεων που ακούσαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Τσούλεϊ. βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, ευκαιρίες ταυτόχρονα και δυνατότητες και η σωστή διακυβέρνηση προσπαθεί να διαρθρώσει ακριβώς ε, τις δυνατότητες αυτές. Πρώτα ερωτήσεις προς τον κύριο Σαστέλ γιατί θα πρέπει να φύγει λίγο νωρίτερα. Η κυρία Ρόιτεβα ερώτηση στον κύριο Σαστέλ και κάποιος άλλος ειδικά για τον κύριο Σαστέλ όποιος έχει ερώτηση. κύριε Γκέπχαρτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Σαστέλ, Αναφερθήκατε στο θέμα της ε, μεταφοράς ε, της οδηγίας για τις υπηρεσίες ε, και τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί. Μας είπατε ότι θα θέλατε η μεταφορά αυτή στην εθνική νομοθεσία να γίνει ταχύτερη. Αυτό έχει σημασία γιατί σε μια τέτοια διαδικασία δικονομική τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αναφερθούν στη μεταφορά αυτή. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για την οδηγία αυτή και η διαδικασία αμοιβαία αναγνώρισης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη και είχα προτείνει μια τριετή μεταβατική περίοδο. Αντίθετα όμως τότε οι υπουργοί επέμειναν στα δύο χρόνια. Και τελικά βλέπω ότι χρειάστηκαν μήνες ολόκληροι για να πετύχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν οι εκπρόσωποι των διαφόρων χωρών να είναι συνυπεύθυνοι στα πλαίσια της νομοθετικής δραστηριότητας και της ταχύτητας μεταφοράς της νομοθεσίας της κοινοτικής. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι η ποιότητα των νομοθετικών αυτών μεταφορών. Το θέμα είναι να μην δουλεύουμε απλά γρήγορα, αλλά να δουλεύουμε σωστά. Γι' αυτό και η πρόταση 47 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να υποστηριχθεί. Πράγματι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο θα επιτρέψει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι οδηγίες στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν και το Συμβούλιο να εκφραστεί και να σταματήσει να κρύβεται. Ευχαριστώ η κυρία Ρούλε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Είχαμε μία διαφωνία προημερών για την έκθεση Βάισκερμπερ και το Συμβούλιο δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει την παραμικρότερη επικοδομητική προσπάθεια και απλά συστηματικά έβαζε εμπόδια στις προσπάθειες των άλλων. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση αν ο πίνακας αυτός δεν λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι στο γενικότερο θέμα. Η ποιότητα της μεταφοράς μιας νομοθετικής ρύθμισης εξαρτάται από την ποιότητα της ίδιας της νομοθετικής ρύθμισης. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την ποιότητα της νομοθετικής μας εργασίας και παραγωγής Σαν παράδειγμα το 2004 είχαμε κάνει μία αναθεώρηση σχετικά με την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες για να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα. Το μόνο που δεν κάναμε είναι να εξυγχρονίσουμε οτιδήποτε. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε σχέση με τα θέματα της ποιότητας. Τελευταίο θέμα, οι προσφυγές επί παραβάση. Οι διαδικασίες αυτές που έχουν πει ότι δεν είναι καθόλου διαφανείς, είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες και γενικά υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά τους. Ο καθηγητής Μόντι έχει κάνει πολύ σωστές προτάσεις. Έχει προτείνει η διαδικασία να μην παρατείνεται πέραν των 6 μηνών ή των 12 μηνών. Αλλά οι προτάσεις του κυρίου Μπαρνιέ δεν το περιλαμβάνουν αυτό. Ελπίζω τα αυτιά που άφησε ο Μπαρνιέ στην αίθουσα να ακούσουν το σχόλιο μου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα το πιο σκοτεινό από τη διαδικασία προσφυγής επί παραβάση εις βάρος των κρατών από πλευράς Επιτροπής. Ρόιτοβα. Ε, εγώ έχω ένα, μια ερώτηση για πολλούς ομιλητές, ε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η δική μου ερώτηση είναι έτσι πιο φιλοσοφική. Ε, είναι σωστό να πούμε ότι τα κράτη-μέλη πιστεύουν πως η εσωτερική αγορά είναι επιτυχημένη και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Πιστεύετε ότι πραγματικά θέλουν την εναρμόνιση κανόνων τα κράτη-μέλη. Δεν πιστεύετε ότι ε, αποσυνθέτουμε πιο πολύ από το να συνθέτουμε. Γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερες προσπάθειες να επιβραδυνθεί εναρμόνιση, να επιβραδυνθεί ολοκλήρωση. Ας δούμε την, τον το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και άλλα θέματα που θα βοηθούσαν και τις επιχειρήσει και τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν την εσωτερική αγορά, την ενιαία αγορά. Και μετά, έχω και άλλη μια ερώτηση για το ψηφιακό περιβάλλον, θα τη θέσω αργότερα. Ευχαριστώ. Δύο ακόμα ερωτήσεις και μετά θα κλείσουμε αυτό το γύρο. Εντάξει κύριε Σαστέλ κυρία Τάιλα και μετά η Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Παρακαλώ σύντομε ερωτήσει. Γιατί ο κ. Σαστέλ θα πρέπει να φύγει. Μπορώ να περιμένω τον επόμενο γύρο γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι για την ψηφιακή οικονομία. Άννα Μαρία. την ερώτηση στον Υπουργό και μου είπε ότι θα μου απαντήσετε εσείς. Μου το υποσχέθηκε. Σας άκουσα να μιλάτε για την μεταγραφή. Συνεπώς ε, χαίρομαι που δίνετε τόση σημασία όσο και εμείς στην ε, μεταγραφή της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, της υφιστάμενης νομοθεσίας. Το ερώτημά μου το εξής. Τι θα κάνετε κατά τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας προκειμένου να ενθαρρύνετε και να υποστηρίξετε τα κράτη-μέλη όχι μόνο στην μεταγραφή αλλά και στην σωστή εφαρμογή Τη υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Εσωτερική Αγορά. Για παράδειγμα, την οδηγία αγαθών, λύσεις μίλησε την οδηγία υπηρεσιών. Ο υπουργό σα μίλησε για το τυρί το οποίο πουλιέται ε, σε, ένα πακέτ, ε, σε πακέτα 40 κιλών στη μία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πακέτα μόνο 15 κιλών σε άλλη. Ε, υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία επιβάλλουν πρόσθετε, πρόσθετους όρους για τα πιστοποιητικά, για πρόσθετες δοκιμές, για, ακόμα και για προϊόντα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στις αγορές. Υπάρχει κατάλογος με τέτοια προϊόντα. Ε, λέτε ότι είναι μια Ευρώπη που ε, ε, οικοδομείται αλλά το αγνοεί. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω μάλλον, μέχρι το τέλος του χρόνου να συγκαλέσετε μια συνάντηση του, του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα σε υπουργικό επίπεδο, γιατί πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του σε υπουργικό επίπεδο για να επανεκκινήσει η εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Α, όχι. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Ωραία. Κυρία Γκεβάρτ, ε, σας ε, ποια ήταν η προσωπική μου άποψη. Ε, δεν είμαι ενθουσιασμένος, είμαι έτσι λίγο, έχω μια ενδιάμεση άποψη. Ε, το Συμβούλιο δεν έχει πάρει θέση, συνεπώς δεν μπορώ να εκφράσω, ε, δεν, μπορώ να εκφράσω την άποψή του. Εγώ πρέπει απλώς να είμαι συνετός στην προσωπική άποψη που εκφράζω. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι απαραίτητη γρήγορη μεταγραφή, αλλά είναι απαραίτητη και η ποιότητα της μεταγραφής. Προσωπικά, ε, στο εσωτερικό της βελικής κυβέρνησης ε, συνεχώς αντιμετωπίζω προβλήματα καθυστερημένης και κακής μεταγραφής και εδώ και αρκετά χρόνια ε, έχω ε, επιχειρώ και έχω καταφέρει η βελγική κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει την ανάγκη γρήγορης και ποιοτική μεταγραφής. Συνεπώς, εξ ονόματος ε, των 27 δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά μπορώ να σας πω ποια είναι η δική μου άποψη και τι κάνω εγώ στη δική μας κυβέρνηση. Ήδη παίρνουμε μέτρα έτσι ώστε η μεταγραφή να επιταχυνθεί και να είναι ποιοτική. Δεν μπορώ όμως να εκφράσω την άποψη των κρατών μελών για αυτό το θέμα. Για την κυρία Ρούλε, είναι αλήθεια ότι αν ο νομοθέτης ε, είχε υπόψη την ανάγκη απλοποίησης της νομοθεσίας, τα κράτη-μέλη ε, θα μετέγραφαν την νομοθεσία αυτή πολύ πιο εύκολα. Σε ό,τι αφορά τη ε, διάρκεια της ε, διαδικασίας και επί παραβάση, ε, ειλικρινά σας λέω ότι ορισμένες φορές, ίσως και πολύ συχνά, ε, οι καθυστερήσει οφείλονται στα κράτη-μέλη, αλλά μερικές φορές οφείλεται και στην Κομισιόν. Οφείλονται και στην Κομισιόν. Γιατί πολλές φορές περιμένουμε τις απαντήσεις της Κομισιόν στα ερωτήματα που εμείς έχουμε θέσει για αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε πολλές φορές και μάλιστα πολύ καιρό τις απαντήσεις κομισιών. Και αυτό δημιουργεί πρόσθετες καθυστέρησεις. Αυτό το λέω προσωπικά, δεν μιλώ εξ ονόματος των κρατών μελών. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία εδώ και τρία χρόνια. Κυρία Ρόιτοβα, Μη λέτε η Προεδρία του Συμβουλίου ή οι διαδοχές Προεδρίες του Συμβουλίου επιβραδύνουν κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την, εσωτερική, με την αγορά. Όχι, μην το λέτε αυτό. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά πόσο μια Προεδρία μπορεί να θέλει να σημειώσει πρόοδο. Έχετε μπροστά σας τους εκπροσώπους της Βελικής Προεδρίας. Το μόνο τομέα το οποίο αναφέρατε της, ε, του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας η δική μας Προεδρία δεν είχε κάνει ποτέ τόσες προσπάθειες ε, ο, καμία άλλη προεδρία δεν είχε κάνει τόσε προσπάθειες όσο εμεί να καταλήξουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη παίζουν στο ίδιο παιχνίδι. Ε, δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο είναι αποτελεσματικό. Συνεπώς, επιτρέπεται να ε, αμφισβητείτε την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου, αλλά μην αμφισβητείτε ε, την επιθυμία και την αποφασιστικότητα μιας συγκεκριμένη Προεδρίας ε, που έχει ε, προσπαθήσει του τελευταίου μήνες όσο οποιαδήποτε άλλη, σε όλα τα επίπεδα, για να περάσει το θέμα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Αύριο το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην έβρεση συμφωνίας. Ελπίζω να καταφέρουμε να τελειώσουμε και με ομοφωνία μάλιστα. Κύριε Κοράτσα το πιο χρήσιμο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν η σύγκριση, καλή σύγκριση των πρακτικών των κρατών μελών μας και αυτό θα το κάνουμε ως Βελική Προεδρία 22-24 Νοεμβρίου. Γιατί πολλά κράτη-μέλη έχουν εργαλεία για την καλή και πετυχημένη μεταγραφή. Ε, πολλά κράτη-μέλη όμως βλέπουν την μεταγραφή από μια οπτική γωνία πολύ περιορισμένη που σχετίζεται με την δική τους χώρα με τη συγκεκριμένη χώρα. Δεν έχουν όμω άποψη για το τι γίνεται αλλού και μάλιστα πολλέ φορέ καλύτερα. Γι' αυτό το λόγο 22 Νοεμβρίου ε, οργανώνουμε την βδομάδα μεταγραφή έτσι ώστε να, δρασ... να ενεργοποιήσουμε ένα πραγματικό μηχανισμό ανταλλαγή καλών πρακτικών. Θα αναφέρω το ερώτημά σα το, το έτοιμά σα ε, να συγκληθεί το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα πριν το τέλο τη Βελική Προεδρία. Θα το αναφέρω στον ε, αρμόδιο Υπουργό. Ευχαριστούμε κύριε Σαστέλ, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εφόσον πρέπει να φύγετε, η Προεδρία απαιτεί να είστε παρόν κατά τη διάρκεια των δικών της συνεδριάσεων. Υπήρξαν και άλλες ερωτήσεις σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές και όλους όσους πήραν μέρος στη συζήτηση. Τι διαχειριστικές προσδοκίες έχουμε γύρω από τα θέματα αυτά, γύρω από τα θέματα επίσης ε, της περί ε, της περιαγωγής γύρω από την τιμολόγηση της περιαγωγής εδώ υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εξελίσσονται και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να ακολουθούμε. Πέντε από τις 50 αυτές προτάσεις έχουν σχέση με την ψηφιακή οικονομία, αλλά παρόλα αυτά στην παρουσίαση που έκανε ο δεύτερος ομιλητής, ο κύριος Τσούλαϊ, Υπάρχει μια κάποια σύγχυση ανάμεσα στους διαφορετικούς τομείς πολιτικής οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. Πώς θα τα συντονίσουμε όλα αυτά. Πώς θα μπορέσουμε να συλλάβουμε την ουσία της προσπάθειας. Και δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τους ε, πολίτες μας και να τους απογοητεύσουμε ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή όπου αντίθετα και συμφωνώ με τον καθηγητή Μόντι ότι τώρα είναι η στιγμή να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό. Είμαστε στο τέλος του 2010. Περνάμε στο 2012 λέει η ομιλήτρια πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει να δείξουμε τι βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε. Και ένα σχόλιο επιπλέον, μιλήσατε για το ανθρώπινο δυναμικό, μιλήσατε για την οικονομία της γνώσης και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Τι περιμένει κανείς από το επιχειρηματικό περιβάλλον, πώς μπορεί να προσαρμοστεί στην οικονομία της γνώσης το άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτεβα συμπληρωματικά. θα ήθελα να σχολιάσω την δεύτερη ομιλία. Πράγματι η εσωτερική αγορά δεν είναι ένα απομονωμένο κλειστό σύστημα. Λειτουργεί στα πλαίσια των ενιαίων αγορών, των σφαιρικών, των παγκοσμιοποιημένων αγορών. Και αυτό επηρεάζει ε, και τα μέτρα τα οποία παίρνουμε στο ψηφιακό περιβάλλον αναφερθήκατε ανάμεσα σε άλλα θέματα ότι αντιμετωπίζουμε αρκετές δυσκολίες. Τις γνωρίζουμε τις δυσκολίες αυτές. Έχουμε μιλήσει για τις δυσκολίες αυτές εδώ και αρκετά χρόνια σε δημόσιες ακροάσεις. Έχουμε επίσης δυσκολίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. η έκθεση που είχε υιοθετηθεί από αυτό το κοινοβούλιο σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον είχαμε ορίσει 25 μέτρα πάνω στα οποία ξεκίνησε να εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαρωτώ με εδώ λοιπόν. Έχετε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες κύριε Τσούλα για μας. σχετικά με τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει στο παρελθόν. Και δεύτερον, και αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό. Η εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο στο διαδίκτυο, με το περιεχόμενο του διαδικτύου. Δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός και αν δεν υπόκειται σε μία εκ των προτέρων σφαιρική συμφωνία γιατί ζούμε σε ένα σφαιρικό περιβάλλον, οι επικοινωνίες λειτουργούν σφαιρικά και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να μην ε, το αγνοούμε. Προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε την εσωτερική αγορά, θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα σύνορα του Σέγγεν, να συζητήσουμε τα θέματα της εναρμόνισης και με τους υπολείπους εταίρους. Κύριε Ρόιτεβα. Θα ήθελα να ρωτήσω από τον κύριο Τσούλε και από τον κύριο Μόντι να δώσουν απαντήσεις. Η κυρία Στάιλερ απευθύνθηκε άμεσα μάλιστα και στον κύριο Μόντι, προς τον κύριο Μόντι. Για την περιαγωγή δεδομένων. Νομίζω ότι τα πράγματα εδώ είναι συμβατά με αυτά που είπε ο κύριος Μόντι. Είναι καιρός κάποιες αυτές τις υποσχέσεις να τις κάνουμε πραγματικότητα γιατί υπάρχουν πολλές προσδοκίες οι πολίτες βλέπουν ποιες είναι οι δυσκολίες του τι συμβαίνει σήμερα όταν ταξιδεύουν, όταν προσπαθούν να κάνουν μια αγορά στα πλαίσια του διαδικτύου σε καθημερινή βάση και όσο καθυστερούμε για τη ρύθμιση αυτών των προβλημάτων θα χάσουν οι πολίτες εμπιστοσύνη στις διαδικασίες τις οποίες χρησιμοποιούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς όλα αυτά μπορούν να γίνουν αντικείμενο συντονισμού. Ελπίζω στο τέλος να υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα συντονισμού. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ε, πρόεδρος Μπαρόσο να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. σχετικά με τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη προτείνει, τι ε, αποτελέσματα έχουμε. Νομίζω ότι για την ενιαία ψηφιακή αγορά βλέπουμε ότι δεν ισχύει το να δημιουργήσουμε μόνο κάποια τμήματα αυτής της αγοράς για να λειτουργήσει. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος ταυτόχρονη σε πολλούς τομείς. Επί της ουσίας βλέπουμε ότι η απόφαση αυτή έχει τεράστια σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Έχουν εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο θα κάνουν πράγματα στο διαδίκτυο καινοτόμα που δεν είχαν κάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς κινδύνους του πακέτου που έχουμε μπροστά μας είναι ότι στην ουσία έχουμε κολλήσει σε κάποιους τομείς που έχουμε συζητήσει και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και δεν σημειώνουμε πρόοδο και αν πραγματικά δεν προχωρήσουμε σε θέματα όπως η προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα των καταναλωτών τότε το πρόβλημα θα είναι πολύ πιο έντονο το επιχειρηματικό περιβάλλον. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους απαιτείται να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο οι μικρομεσαίες περνούν όλο και περισσότερο στο δικτυακό κόσμο. Απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια λοιπόν, απαιτείται να προχωρήσουμε στον τομέα των ηλεκτρονικών υπογραφών, στο λεγόμενο invoicing στην έκδοση τιμολογίων. Υπάρχουν και άλλοι τομείς πολύ πιο δύσκολοι όπως η φορολογία. Αν δούμε τι γίνεται με τα διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ σαν παράδειγμα, απαιτείται να υπάρξει πρόοδος και στους τομείς αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ για όλη την Ευρώπη αλλά απαιτείται να υπάρξει πρόοδος σε σχέση με την εφαρμογή κάποιων από, αυτών, από αυτές τις αρχές. Γύρω από την σφαιρική φύση του διαδικτύου πράγματι το διαδίκτυο λειτουργεί παγκόσμια σφαιρικά και θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος και σε διεθνές επίπεδο. Δεν νομίζω όμως το να υπάρξει πρόοδος σε διεθνές επίπεδο ότι είναι προϋπόθεση για να υπάρξει πρόοδος σε ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Όταν εξετάζουμε σαν παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές στρέφονται στο ίντερνετ, προφανώς θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν κάποιες διεθνείς συμφωνίες προστασίας των καταναλωτών. Τη απουσία όμως αυτών των συμφωνιών είναι κατανοητό οι καταναλωτές να βλέπουν τις διαφορές προστασίες που έχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο όπου υπάρχει πολύ μικρότερη δυνατότητα διακανονισμού θα έλεγα της συναλλαγής. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο καταναλωτής είναι οι διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες της Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καθηγητής Μόντι θα θέλει και αυτός να σχολιάσει. Σας ευχαριστώ πολύ που επιμένετε τόσο ευγενικά. Να πω απλώς ότι ε, άκουσα δύο έννοιες με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα. Πρώτον, καλύτερη ορατότητα και συνεκτικότητα σε μια ολιστική προσέγγιση, πράγμα το οποίο σημαίνει και μεγαλύτερος ρόλος για τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Δεύτερον, όπως είπε ο κύριος Ζούλεγκ, σαφώς να γίνει η διαβούλευση η τετράμινη, αλλά παράλληλα οι υπεύθυνε αρχές να συνεχίζουν να προσπαθούν να βρουν μία συμφωνία, μία αρχή συμφωνίας, συνένεσης, συμβιβασμού μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών και μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε επιτυχώς να ολοκληρώσουμε και τη διαβούλευση. Πρόεδρος, ένα ναι μόνο μπορώ να πω σε αυτό το οποίο προτείνατε κύριε Μόντι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτού του πάνερ Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και όλους αυτούς οι οποίοι έθεσαν ερωτήσεις. Έλαβα και μια γραπτή ερώτηση από τον κύριο Μπέρντ Σμίτλερ για, για τα εμπόδια, τα προστατευτικά στον τομέα των βιοκαυσίμων και για έναν ειδικό φόρο για την ε, ενέργεια, για τον τομέα της ενέργειας, Απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ερώτηση αυτή. Δεν έχουμε κανέναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πάνελ. Έχουμε όμως εκπρόσωπο του DigiMarkt μαζί μας. Επομένως θα μεταβιβάσω την ερώτηση αυτή στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα προωθηθεί στον αρμόδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η ερώτηση. Περνάμε στο επόμενο πάνελ επικεφαλής του οποίου είναι ο κύριος Κρίστιαν Μπουζόη και θέμα του τελευταίου αυτού πάνελ είναι η επικοινωνία και ενίσχυση των πολιτών στα πλαίσια της ε, ενίας αγοράς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάποια εισαγωγικά σχόλια. Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίτευγμα για το οποίο μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι. Ένα επίτευγμα με πάρα πολλές δυνατότητες για τους, πολ... πολίτες και τις επιχειρήσεις και λυπάμαι που ένα μεγάλο τμήμα της ενιαίας αγοράς δεν το έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί. Μόλον ότι υπάρχουν πολλά πλέον εκτήματα, η υποστήριξη του πολίτη για την ενιαία αγορά δεν ήταν πάντα όσο δυνατή θα έπρεπε να είναι και η κατάσταση δεν βελτιώνεται σήμερα με την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Προκειμένου να τροποποιηθούν τα πράγματα θα πρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς την ενιαία αγορά προκειμένου να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε και ένα υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης του πολίτη. Πρέπει να βρούμε καλύτερες λύσεις προκειμένου να οικοδομήσουμε μια ενιαία αγορά η οποία να βρίσκεται όσο δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Μία ενιαία αγορά λοιπόν, η οποία συνεχώς θα φέρει τη θέμενη αξία για τους πολίτες. Μία ενιαία αγορά η οποία αποτελεσματικά θα αποκρίνεται στι ανάγκε του πολίτη και που θα βελτιώνει τη ζωή του πολίτη. Οι εκπρόσωποι των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι οι πλέον αρμόδιοι για να μας πούνε ποιες είναι οι απαιτήσει και προσδοκίες των πολιτών από την ενιαία αγορά. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να μιλήσω για το ζήτημα αυτό της επικοινωνίας και της ενίσχυσης των πολιτών με την κυρία Μονίκ Γκογιάνς, Γενική Διευθύντρια της ΜΠΕΟΚ, που είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός εκπροσώπης των καταναλωτών, και με τον κύριο Φιλίπ Ντεμπούκ, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Business Europe. Πρωτού δώσω το λόγο, θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία σημαντικά σημεία στη συζήτηση αυτή. Η πράξη για την ενιαία αγορά, την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Οκτωβρίου, περιέχει κάποιες προτάσεις για την ενίσχυση των πολιτών. Ορισμένες από τις προτάσεις αυτές βασίζονται σε συζητήσεις και σε ιδέες που έχει υποβάλει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα αποτελέσει πλέον την μοναδική ενιαία θηρίδα για την εξυπηρέτηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό σε, σχέση με τα, σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένε προτάσεις που γίνανε για να επιληθούν επιμέρους προβλήματα αποτελούν πραγματική πρόοδο και βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτών και επιχειρήσεων. Μια σημαντική πρόταση της πράξης της ενιαίας αγοράς έχει να κάνει με την επίλυση των προβλημάτων και συγκεκριμένα μέσω του Solvit. Δίκτυο το οποίο με απασχόλησε και που θεωρώ ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών. Αν θέλουμε πραγματικά τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίδει η ενιαία αγορά, η ενιαία αγορά πλήρως, θα πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη που έχουν σε αυτή την ενιαία αγορά. Και θα πρέπει ο μηχανισμός αυτός να είναι άμεσα διαθέσιμος αυτούς. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα για το Solvit. Μολονότι έχει μια πρώτη σημαντική επιτυχία, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα προσωπικού και κάποια νομικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Ελπίζω ότι ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τους εκπροσώπους των πολιτών και των επιχειρήσεων θα καταφέρουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στους τομείς αυτούς. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συνδεθούν περισσότερο συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι εκπρόσωποι των πολιτών και των επιχειρήσεων στην όλη διαδικασία εφαρμογής. Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσει ένας διάλογος με όλους αυτούς τους φορείς πριν την εφαρμογή της πράξης για την ενιαία αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται πλήρω υπόψη οι απόψει του και κατά αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή πολιτική θα αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία για του πολίτε. Αναφέρθηκα σε τρία σημαντικά σημεία, τρεις πρώτες ιδέες, τις οποίες θα ήθελα να θέσω στα πλαίσια της συζήτησης. Πρέπει να βρούμε όμως τους συγκεκριμένου τρόπους με τους οποίους θα καταφέρουμε να φέρουμε την ενιαία αγορά πιο κοντά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την κυρία Μονίκ Γκογένς να μας κάνει τη δική της παρουσίαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Γκογένς. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μάλκομ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκάλεσες για να μιλήσω περισσότερο για τους καταναλωτές στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς και πιο συγκεκριμένα της πράξης για την ενιαία αγορά. Χαιρετίζουμε τη διοργάνωση του φόρουμ αυτού και ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι θα γίνεται πλέον συστηματικά και ότι του χρόνου θα γίνει στην Πολωνία. Χαιρετίζουμε σαφώς λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να υποστηριχθεί. Ενδεχομένως κάποια προκατακτικά σχόλια προτού μιλήσω για την πράξη για την ενιαία αγορά. Στην πράξη για την ενιαία αγορά, όπως και σε πάρα πολλές συζητήσει, υπάρχει μια διαλειτουργικότητα όσον αφορά τους πολίτες και τους καταναλωτές. Θεωρούμε ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση. Σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπώ τα συμφέροντα των πολιτών. Εκπροσωπώ τα συμφέροντα των καταναλωτών, όντας επικεφαλής μιας Ένωσης Καταναλωτών Ευρωπαϊκής. Η εκπροσώπηση του καταναλωτή δεν συνάδει απόλυτα με την εκπροσώπηση ενός ανθρωπίνου όντως. Ο καρδιναλωτής είναι, μια ιδιότητα η οποία παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυθαίρετα τους δύο αυτούς όρους πολίτη και καταναλωτή, γιατί η έννοια είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Αν δούμε τώρα την πράξη για την ενιαία αγορά, στην ουσία τη βλέπουμε. Ακούσαμε τον κύριο Μόντι, ο οποίος πιστεύει ότι θα πρέπει η διαβούλευση να προχωρήσει πολύ γρήγορα, ενδεχομένως και να ολοκληρωθεί σύντομα. Συμφωνώ με την προσέγγισή σας, ενδεχομένως να πρέπει να συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Ωστόσο βρισκόμαστε και στο τέλος μιας διαδικασία που ξεκίνησε από την δέσμευση του κυρίου Μπαρόζο στη νέα του αυτή θητεία που είπε ότι θα πρέπει ο πολίτης πλέον να μπει στην καρδιά της νέας αγοράς. Έχουμε επίσης και την έκθεση του κυρίου Μόντι η οποία υιοθετεί πολλές πρωτοβουλίες φιλικές προς τον καταναλωτή. Και τέλος έχουμε και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον κύριο Γκρέκ. Στην έκθεση αυτή γίνεται μια δήλωση η οποία θέτει πραγματικά τον πύχη στο σωστό επίπεδο. Λέγεται ότι η ευημερία του καταναλωτή θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενιαία αγορά. Η δήλωση πραγματικά αυτή θα πρέπει να αποτελέσει το μέτρο αξιολόγηση τη πράξη για την ενιαία αγορά είναι ικανή η πράξη και η αγορά να ανταποκριθεί στη δήλωση αυτή. Δεν θα ήθελα να με παρεξηγήσετε. Έχω λίγα λεπτά μόνο στη διάθεσή μου, επομένω δεν θα καταφέρω να επισέλθω σε όλε τι λεπτομέρειε που είναι σημαντικέ για έναν καταναλωτή για την ενιαία αγορά. Είδαμε ότι είχε καταβληθεί τεράστια προσπάθεια, ιδίω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπήρξε μια πολύ σημαντική διοργανική και διυπηρεσιακή συνεργασία και διαβούλευση και σαφώ έχουν επιτευχθεί πολλά πράγματα. Δικό μου όμω ρόλο είναι να δείξω επικριτική στάση και θα ήθελα να σα δείξω ποια είναι η σκοπιά του καταναλωτή για τα έχουν προταθεί μέχρι στιγμή έχουμε λοιπόν επιτάπητο. Θεωρούμε σαφώς ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσε πρωτοβουλίες και θα επανέλθουμε σε αυτέ. Θεωρούμε όμω να έχει δοθεί απαραίτητη προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες εκείνες που δυνάμει μπορούν να έχουν θετική επίπτωση στην ευημερία του Ευρωπαίου καταναλωτή. Και υπάρχει μία ακόμα ανησυχία. Είναι πολλές οι περιστάσεις εκείνες στις οποίες αντιμετωπίζουμε την ενιαία αγορά ως μία απλή διασυνοριακή δραστηριότητα για τους καταναλωτές. Κοιτάξτε, και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις η ενιαία αγορά θα πρέπει να σημαίνει ένα ισότιμο επίπεδο δραστηριότητας, είτε πρόκειται για εθνικές δραστηριότητες, είτε πρόκειται για διασυνοριακές δραστηριότητες, είτε είναι κανείς ενεργός ή παθητικός καταναλωτής. Το να υποτιμούμε την ενιαία αγορά προσεγγίζοντάς την μόνο ως μία διασυνοριακή συναλλαγή, είναι κάτι που δεν τιμά καθόλου το όλο εγχείρημα το 95% των δραστηριοτήτων στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς είναι εθνικές δραστηριότητες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αναφερόμαστε και να επικεντρωνόμαστε μόνο στις συνοριακές δραστηριότητες και αυτές οι συνοριακές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν μια προσθέμενη αξία. Δεν πρόκειται ποτέ να πάω να αγοράσω σε μια άλλη χώρα το ψωμί μου, εκτός και αν μένω βέβαια κοντά στα σύνορα. Επίσης, η πράξη για την ενιαία αγορά κάνει μια κατηγοριοποίηση των προτάσεων. Νούμερο 1 την είναι καλό για τις επιχειρήσεις, νούμερο 2 την είναι καλό για τους εργαζομένους, νούμερο 3 την είναι καλό για τις διαδικτυακές ε, υπηρεσίες και στο τέλος βλέπουμε κάποια στιγμή και τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα για τους ε, καταναλωτές. Πιστεύω ότι θα πρέπει η προσέγγιση να είναι ολιστική και σφαιρική σε κάθε επίπεδο. Κάθε φορά που μιλάμε για τα δικαιώματα του δημιουργού ή για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Βρεσιτεχνία, θα πρέπει να γνωρίζουμε ταυτόχρονα τι είναι καλό για τον ίδιο τον παραγωγό, τι είναι καλό για τον ίδιο τον επιχειρηματία και τι είναι ωφέλιμο όμω και για τον ίδιο τον καταναλωτή. Πρέπει να υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση σε όλε τι προτάσει. Και συμφωνώ με τον κύριο Μόντι, ο οποίο είπε Α σταματήσουμε επιτέλου διαβουλεύσει και προχωρήσουμε στη δράση υπάρχουν πολλές προτάσεις της πράξης για την ενιαία αγορά που είναι ουσιαστικά προτάσεις που έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Ορισμένες προτάσεις έχουμε δει πριν από κάποιες δεκαετίες μάλιστα θα σας έλεγα. Ε, έχει έρθει λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσουν τα λόγια και να περάσουμε στις πράξεις. Ας αναφερθούμε τώρα στα πιο σημαντικά σημεία, στις πιο σημαντικέ προτεραιότητες για το καταναλωτή που υπάρχουν βέβαια στην πράξη για την νέα αγορά. Ένα αισιόδοξο βέβαια θα έλεγε ότι πάλι καλά που ο καταναλωτή βρίσκεται στην πράξη για την ενιαία αγορά. Δεν αρκεί όμω αυτό. Α είμαστε και λίγο πιο ρεαλιστέ. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο φιλοδοξία. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βαν Κουίκεμποργκ. Είπε την ουσία των πραγμάτων. Στο τέλος βλέπετε ότι ε, αν φύγουν κάποια στοιχεία, τι θα παραμείνει από την πρόταση αυτή αν εξαλειφθούν τα προβληματικά στοιχεία, τι πρόκειται να παραμείνει. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι σε σχέση με την εφαρμογή των προτάσεών μας. Καταρχάς, συλλογικές αποζημιώσεις. Ακούσαμε την κυρία Γκέπχαρτ, αναφέρθηκε ήδη σε αυτό. Δεν υπάρχουν τα ίδια μηνύματα στα αυτά τα δύο έγγραφα. Πρέπει να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς θέλετε. Αυτή είναι η πρόταση, αν θέλετε να πουλήσετε ακριβώς την ενιαία αγορά στους καταναλωτές. Πολλά έχουν υποθεί σε σχέση με το ADR, ADR in order to uh, solve disputes, έτσι ώστε να λύνονται τα προβλήματα και οι διαφορές που δημιουργούνται στα πλαίσια της κατανάλωσης. Είχαν ξεκινήσει πρωτοβουλίες σχετικά με το ADR εδώ και 12 χρόνια, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα είτε σε εσωτερικό επίπεδο είτε σε διαμεθοριακό επίπεδο με ελάχιστες τομεακές εξαιρέσεις. Ας πούμε πιστοτικές υπηρεσίες, διαμεθοριακές πιστοτικές υπηρεσίες, αφού δεν υπάρχει αγορά διαμεθοριακή, γιατί να υπάρχει ADR. Ε, ε, ε, ας φτιάξετε πρώτα την αγορά και μετά φτιάχνετε το σύστημα αυτό. Ο τρόπος των συλλογικών αποζημιώσεων αντιμετωπίζεται ε, με πολύ διπλωματικό τρόπο και αυτό δείχνει σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να αποκωδικοποιήσουν την γλώσσα αυτή ότι έχει παγώσει η πολιτική βούληση να προχωρήσουν. Οι προηγούμενοι ομιλητές ε, αναφέρθηκαν σε πολλά από αυτά τα θέματα αλλά όλοι πιστεύουν ότι αυτές οι συλλογικές αποζημιώσεις δεν θα πρέπει να τις ονοματίσουμε. Υπάρχει φόβος να εμπλακούμε και ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται στην ενιαία πράξη δεν δείχνει ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα στους καταναλωτές να μπορούν να προσφεύγουν συλλογικά στα δικαστήρια είτε ε, στις ε, εθνικές είτε στις κοινοτικές ε, αρχές. Ο κύριος Μπαρνιέ αναφέρθηκε στην πρόταση αυτή σχετικά και με το θέμα της εναλλακτική επίλυσης διαφορών. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα πάντως συλλογικών αποζημιώσεων και συλλογικών προσφυγών πολύ πιο πλήρες από το τωρινό. We is on Επίσης το θέμα των νομικών διαφορών σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Αυτή η πολυδιάσπαση νομική δημιουργεί προβλήματα. Η ασφάλεια των πληρωμών, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, ε, τα προϊόντα θα παραδοθούν. Υπάρχουν ανησυχίες από τους καταναλωτές και δεν είναι μόνο θέμα διαμεθοριακού εμπορίου, διασυνοριακού αν θέλετε εμπορίου. Είναι και θέμα εθνικού εμπορίου πολλές φορές, εσωτερικού εμπορίου. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι προτάσεις που θα γίνουν στη συγκεκριμένη οδηγία που είναι υποσυζήτηση θα δώσουν κάποιες λύσεις θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στις, στα δικαιώματα του δημιουργού και στα δικαιώματα του χρήστη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν θέλουμε να είναι ενημερωμένοι και ισχυροί οι καταναλωτές, θα πρέπει να υπάρχουν μέσα για τον έλεγχο των αγορών και να δούμε πού υπάρχουν εγγυήσει για τους καταναλωτές. Οι διαδικασίες μελέτης επιπτώσεων έτσι όπως έχει ανακοινωθεί θα καλύψουν και τον κοινωνικό τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και σίγουρα θα είναι ένα επιπλέον μέσο για περισσότερη διαφάνεια όταν τεθεί σε πρακτική. Θέλουμε μεγαλύτερη εμπλοκή επίσης και των οργανώσεων των καταναλωτών να εντοπίσουμε σωστά τους δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και στα πλαίσια της ε, ανείχνευσης των βασικών προβλημάτων, των 20 βασικών προβλημάτων όπως λέει και η έκθεση Γκρέφ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια τακτική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς βαθίζει η ενιαία αγορά για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Και αυτό μας οδηγεί τώρα σε ένα τελευταίο και γενικό θέμα. Όλοι μιλάνε για το κεντρικό ρόλο του καταναλωτή στην ενιαία αγορά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδέα για το τι θέλει κανείς σαν πολιτικός να είναι η πολιτική για την κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σέβομαι όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται στα διάφορα θεσμικά όργανα. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει έλλειψη πολιτικού οράματος για το τι θέλουμε η προστασία του καταναλωτή να είναι. Το έχουμε παρατηρήσει αυτό και σε σχέση με τις συζητήσεις που έχουν γίνει για την προστασία του καταναλωτή, εναρμόνιση, ελάχιστη εναρμόνιση ε, και πάρα πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες δείχνουν ότι η ευημερία σε εισαγωγικά των καταναλωτή θεωρείται ότι είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα της κατάργησης των εμποδίων για το εμπόριο. Εγώ δεν θα ήθελα να θεωρείται σαν κάτι το δευτερεύον η προστασία του καταναλωτή. Θέλουμε να είναι στόχος βασικός. Αυτοί που ασκούν με την πολιτική πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτό και θεωρούμε πάρα πολύ θετικό αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόταση και στην πρόταση μάλιστα του κυρίου Μπαρνιέ, αυτή η νέα επιθυμία και βούληση πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη εμπλοκή εταίρων εκτός του επιχειρηματικού κόσμου, δηλαδή ομάδων εμπειρογνωμόνων, καταναλωτών κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και ακούγεται από τότε που ανέλαβε ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Αυτό ε, χρειάζεται, είναι προαπαιτούμενο. Θέλουμε να γίνει. Αλλά αυτό σημαίνει βέβαια και ισχυρές οργανώσεις καταναλωτών. που να έχουν αρκετούς πόρους και εμπειρογνωσύνη, εμπειρογνωμοσύνη στην ε, διάθεσή τους. Έχει σημασία αυτή η τελευταία παρατήρηση. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα. Τι συμβαίνει σήμερα. Βλέπουμε ότι τον τελευταίο μήνα μάλιστα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη πολλές οργανώσεις καταναλωτών στην ουσία βλέπουμε ότι συρρυκνώνονται οι αρμοδιότητές τους από τις κυβερνήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Το ίδιο γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι προϋπολογισμοί αυτών των καταναλωτικών οργανώσεων αμειώνονται συνεχώς και κάποιες απειλούνται με εξαφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Consumer Focus που είναι η βασική οργάνωση και δημιουργήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια, απειλείται με κατάργηση. Η ανάλυση την οποία κάνω εγώ και είμαι λίγο προκλητική ίσως, είναι ότι πράγματι έχει υπάρξει μια κακή διαχείριση του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει υπάρξει μια οικονομική κρίση, οι κυβερνήσεις υποστήριξαν τις τράπεζες, καλά κάνανε ίσως, για να αποφύγουμε τα χειρότερα σενάρια. Οι τράπεζες πάνε πολύ καλύτερα τώρα και έχουν κέρδη. Κάποιοι traders ε, ή πήραν μπόνους ε, τα τελευταίο χρόνο που συνολικά ε, τα μπόνους τους μόνος είναι πιο ψηλά από τη συνολική ετήσια αμοιβή των εργαζομένων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, για να είμαι πιο συνοπτική. Οι τράπεζες συμπεριφέρθηκαν άσχημα και γι' αυτό τιμωρούνται οι οργανώσεις των καταναλωτών. Τώρα τι πολιτικό μήνυμα είναι αυτό το οποίο στέλνετε στους καταναλωτές και τους πολίτες κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Και αναρωτιέστε γιατί η ενιαία αγορά δεν είναι ελκυστική για τους πολίτες. Λοιπόν, ίσως κάτι πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα και αυτό θα το θεωρούσαμε κάτι το θετικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκόγενς. Καλό τώρα τον κύριο Φιλίπ Ντεμπούκ να πάρει το λόγο. Είναι Γενικός Γραμματέας της Business Europe. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του πάνελ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας αυτή, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να τοποθετηθώ ως εκπρόσωπος των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την ε, πράξη για την ενιαία αγορά. Θεωρώ ότι η παρέμβαση μου αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή, γιατί ακούσαμε πρώτα την παρουσίαση για την πράξη για την ενιαία αγορά. Είχα όμω και εμείς τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην Επιτροπή εκείνη, η οποία συζήτησε, στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς του Κοινοβουλίου, που συζήτησε την έκθεση του κύριου Γκρέχτ. Και χαίρομαι πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να έχω μια ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Γκόγιένσα, εκπρόσωπο τη ΜΠΕΚ. Δεν το είπε, αλλά συνεργαζόμαστε για κάποια ζητήματα και πρέπει να πω και με επιτυχία. Σε αντίθεση βέβαια με τον Μάριο Μόντι, εγώ πολλές φορές καλούμε να αντισταθώ στις πολύ ευγενικές προσκλήσεις που μου κάνει για διάφορα ζητήματα. Πάντως στους περισσότερους τομείς καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε. Και εδώ υπάρχει και μία παρανόηση την οποία θα ήθελα να διαλευκάνω κατά κάποιο τρόπο. Η ενιαία αγορά δεν είναι μόνο ένα οικονομικό σχέδιο, δεν είναι ένα σχέδιο που προορίζεται μόνο για τις επιχειρήσεις. Είναι και το είπε, το υπογράμμισε η κυρία Γκογένς και το έχουν υπογραμμίσει και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι θετικό και για τους εργαζόμενους και για τους καταναλωτές. Προκειμένου όμως να έχουμε μία ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν μία εσωτερική αγορά η οποία να υπερβαίνει την εθνική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνα στην οικονομία και δεν θα ήθελα βέβαια να τοποθετικό αυτόν τον τρόπο μπροστά από ένα καθηγητή, τον κύριο Μόντι. Πάντω το μέγεθο των επιχειρήσεων εξαρτάται αναλογικά από το μέγεθο τη εγχώρια αγορά, τη εθνική αγορά. Προέρχομαι από το Βέλγιο και γνωρίζω πολύ καλά το ζήτημα αυτό και πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Το μέγεθος των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι τέτοιο που να τους επιτρέπει να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Και γι' αυτό, για όλους αυτούς τους λόγους, ως Business Europe Είμαστε 100% υποστηρικτές της έννοιας της ενιαίας αγοράς και υποστηρίζουμε πλήρως την πράξη για την ενιαία αγορά. Σαφώς υπάρχουν δυσκολίες, σαφώς αντιστεκόμαστε σε κάποιες από τις προτάσεις που έχουν γίνει, υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί, αλλά εν γέννη υποστηρίζουμε την πρόταση αυτή. Δεν θα ήθελα να επισέλθω αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειε και αριθμητικά δεδομένα. Ακούσαμε πάρα πολλέ λεπτομέρειε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση και σα ζητώ συγγνώμη που πήρα το λόγο τόσο καθυστερημένα. Υπάρχουν πάντω πολλοί ομιλητέ και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι με κάλυψαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όπω είπατε πολλοί, πρέπει να δούμε αν έχουμε τον απαραίτητο την πολυτέλεια του χρόνου για να ασχοληθούμε με τη διαβούλευση. Εμείς τοποθετηθήκαμε για το ζήτημα αυτό και στο παρελθόν συμμετείχαμε σε πολλές διαβουλεύσεις αν αυτές είναι απαραίτητε για πολιτικούς λόγους τότε να συμμετέχουμε και στις μελλοντικέ. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε απτά αποτελέσματα στο τέλος της διαδικασίας διαβούλευσης. Εμείς ως επιχειρήσεις, ως εργαζόμενοι, ως καταναλωτές θέλουμε να δούμε μία πραγματική αισθητή θετική διαφορά ανάμεσα στο πριν και το μετά. Αυτό αποτελεί πραγματική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να, κάνει σωστές προτάσεις και αποτελεί όμως πρόκληση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο και για όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των νομοθετημάτων. Όλοι αυτοί θα πρέπει να συμμετέχουν στη συζήτηση που γίνεται για την ενιαία αγορά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο γιατί πιέζει ο χρόνος να αναφερθώ σύντομα σε κάποια σημεία. Πρώτον, όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Μια θεμελιώδη βελτίωση της διαχείριση της ενιαίας αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφεύγουν κάθε φορά που υπάρχει μια ανησυχία, κάθε φορά που προκύπτει μια διαφορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια πραγματικά ολοκληρωμένη στρατηγική. Ένα Ευρωβουλευτή το είπε πριν από λίγο. Ακούγονται πολλέ διαφορετικέ προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλε αλληλοσυνδέονται με τον ένα τον άλλο τρόπο και έχουν σχέση με την έννοια αγορά προφανώ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση του, να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η εφαρμογή των κανόνων επίση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τρίτον, χρειαζόμαστε μια καλύτερη ρύθμιση και όπως είπε και ο Επίτροπος χρειαζόμαστε το περίφημο smart regulation, της ε, ευφυείς ρυθμίσεις. Τώρα, αντίκτυπος επιπτώσεων. Σαφώς θα πρέπει να λάβει χώρα. Πολλά πράγματα πρέπει να εξεταστούν. Αλλά ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις για την ενιαία αγορά. Ποια είναι τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της πρότασης. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από την αρχή. Και τέλος, Ξέρετε ότι κάθε φορά που εκπροσωπεί κάποιο επιχειρήσει στην Ευρώπη, εκπροσωπεί ουσιαστικά μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Και στόχο μα είναι να διευκολύνουμε την καθημερινή τους λειτουργία μέσω των προτάσεων. Η Μονίκ Γκογέν πριν από λίγο είπε ότι η ενιαία αγορά δεν είναι μόνο διασυνοριακέ συναλλαγές αλλά κυρίω εθνικέ συναλλαγές. Από επιχειρηματική πλευρά, αυτό που θέλω να πω δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο καμία διαφορά. Χρησιμοποιούμε σε 16 χώρε πλέον το ευρώ. Ξεχνάμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλο νόμισμα όταν πηγαίνουμε εκτός της ε, ζώνης του ευρώ. Ακριβώς την ε, ίδια αίσθηση θα πρέπει να έχουμε επιχειρήσεις και καταναλωτές για την ενιαία αγορά. Τώρα, πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο στην εφαρμογή των κανόνων, στην επιβολή των κανόνων. Θεματοφύλακα άλλωστε των συνθήκων είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και τις αποφάσεις του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο όπου επιλύονται κάποια προβλήματα, αλλά πηγαίνει κανείς στο δικαστήριο όταν έχει αποτύχει ουσιαστικά η διαδικασία επιβολής και εφαρμογής. Θα πρέπει οι διαδικασίε σε παραβάση να παρακολουθούνται εκ του και θα πρέπει το όλο σύστημα συμμόρφωσης να είναι αποτελεσματικό. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρχει εδώ καλή συνεργασία να ειμαστε κράτη-μέλη. Και να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με τις μεθόδους αποζημίωσης και προσφυγής. Το ζήτημα αυτό το συζητήσαμε εκτενέστατα. Είμαστε υπέρ του συστήματος εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αποτελεσματικό και ιδιαίτερα φιλικό προς τους καταναλωτές και είναι ένα σύστημα το οποίο είναι λιγότερο δαπανηρό για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Είναι οικονομικά αποδοτικό αν θέλετε το εναλλακτικό αυτό σύστημα επίλυσης των διαφορών. Ξέρετε ότι είμαστε κατά των συλλογικών προσφυγών και αποζημιώσεων. Όχι γιατί μας ενοχλεί το ενδεχόμενο των συλλογικών αυτών προσφυγών, αλλά γιατί φοβόμαστε ότι αντιβαίνει στις προτάσεις που γίνονται στην πράξη και την ενία αγορά. Και το τελευταίο πράγμα που θέλει, που θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι τέτοιο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν στι Ηνωμένε Πολιτείε, συζήτησα το ζήτημα αυτό με του ομολόγου μου εκεί και μου είπαν και αυτοί ότι και αυτοί θα ήθελαν να σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα αυτού των συλλογικών προσφυγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Solvit στη συνέχεια. Πιστεύουμε ότι είναι ένα σύστημα, ένα δίκτυο το οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί ενδεχομένω να πρέπει να το διαφημίσουμε λίγο περισσότερο. ενδεχομένω οργανώσαν αυτέ αυτές που εκπροσωπώ εγώ να πρέπει σε εθνικό και τοπικό επίπεδο να μιλήσουν λίγο περισσότερο για το Solvit και να ενημερώσουν τον πολίτη και τι επιχειρήσει. Σαφώς υπάρχουν επίσης κάποια εμπόδια ακόμα στην ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια τα οποία αντιστοιχούν σε δισεκατομμύρια ευρώ. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα εφίσταται. Το πρόβλημα τώρα είναι το ακόλουθο μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά με την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι υπηρεσίες αποτελούν το 70% του μέσου ΑΕΠ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες θα πρέπει να επιληθούν όλα τα υφιστάμενα προβλήματα των υπηρεσιών μέσω της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Και καταλαβαίνετε ότι εμείς ως Business Europe αλλά και το Eurochamber υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες. Ενία αγορά για τα προϊόντα. Τομέα στον οποίο είχε σημειωθεί σαφώς πρόοδος στο παρελθόν, αλλά όπως είπαν και κάποιοι ευρωβουλευτές σήμερα το απόγευμα, ακόμα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος. Υπάρχουν δηλαδή πολλά μικροπροβλήματα εδώ και εκεί, αλλά αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ενία αγορά. Επίσης, πώς θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε περισσότερο τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε το καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέο νομοθέτημα και ελπίζω ότι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα αυτή η Βελγική Προεδρία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέσο ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έρχομαι στο τέλος, σιγά σιγά. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις καινοτομίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Άκουσα αυτά που είπατε για την ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία, άκουσα αυτά που είπε η βελγική κυβέρνηση, είμαι Βέλγος, τους υποστηρίζω. Πρέπει να κλείσει το θέμα αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε αποδείξει επαρκώς τα πλεονεκτήματα ύπαρξης αυτής της ευρωπαϊκής ευρεσιτεχνίας. Δεν θα είναι τέλεια, αλλά θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Ακούστηκαν επίσης πολλά σημαντικά και για την ενιαία ψηφιακή αγορά και αυτό είναι μείζον θέμα και στα πλαίσια γενικότερα της βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης, όχι μόνο σε επίπεδο λογισμικού αλλά και σε επίπεδο λογιστικού. Εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την, τον, την καταπολέμηση του, του ψηφιακού αποκλεισμού, εν πάση περιπτώσει κτλ. Ένα έκτο θέμα Υπάρχει ένα θέμα σχετικά με την κοινωνική διάσταση της ενίας αγοράς. Και είμαι ευγνώμων προς τον Μάριο Μόντι γιατί είδατε στην έκθεση του ότι κάνει μια προσπάθεια να φέρει σε επαφή όλους τους εταίρους έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε την ένταξη της κοινωνικής διάστασης. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει επίσης στο παρελθόν. Ελπίζω να έχουμε περισσότερες δυνατότητες στο μέλλον εμείς που έχουμε να κάνουμε με την οδηγία για την τοποθέτηση των εργαζομένων προσπαθούμε να βρούμε τους σωστούς τρόπους για την σωστή ενημέρωση των εργαζομένων και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη αναθεώρησης των συνθήκων ε, των εργαζομένων στα πλαίσια, εκτός μάλλον των πλαισίων της συγκεκριμένης οδηγίας. Και ένα δεύτερο θέμα που αφορά πάντα την κοινωνική ε, ρήτρα. Έχουμε ξεχάσει ότι από τη συνθήκη της Λισαβόνας η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι δεσμευτική πλέον και όλα τα στοιχεία πλέον υπάρχουν για συλλογικές ε, προσφυγές και τα λοιπά και ε, απεργίες. Εγώ δεν είμαι υπέρ των απεργιών και προφανώς προσπαθούμε να τις αποφύγουμε. Ένα τελευταίο θέμα αφορά την διεθνή διάσταση της ενιαίας πράξης. Της ενιαίας αγοράς, Η ενιαία αγορά έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο για το ξεπέρασμα της κρίσης και για να αποφύγουμε έντονες προστατευτικές πρακτικές και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ταυτόχρονα όμως η ενιαία αγορά προσφέρει και μια τεράστια πλατφόρμα για αυτούς που έρχονται στην ενιαία αγορά. Όχι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις εισαγωγές, αλλά θα πρέπει να τοποθετούμε τα προϊόντα αυτά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός δίκαιος και να γίνονται σεβαστές όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας για τα εισαγόμενα. Λοιπόν, είμαστε υπέρ των προτάσεων αυτών, είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε τις προτάσεις αυτές, αλλά έχουμε μεγάλη ανάγκη να εφαρμοστούν όλες αυτές οι προτάσεις γρήγορα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Ντεμπούχ. Αγαπητά μέλη, ακούσαμε τη φωνή των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και βλέπουμε ότι υπάρχει μια θετική αντίληψη γύρω από τα θέματα αυτά σχετικά με την ενημέρωση και ενίσχυση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν μπορείτε μέσα σε ένα λεπτό να θέσετε ερωτήσεις προς τους συναδέλφους μου, από τους συναδέλφους μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν όχι, θα δώσω το λόγο μία ερώτηση από πλευράς της Ένωσης Πολωνών Καταναλωτών στην κυρία Γκόιενς και θα δώσουν γραπτή απάντηση. Σας ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Χάρμπορ, τον πρόεδρο της Επιτροπής να κλείσει τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους σας που πήρατε μέρος και που μείνατε, ιδιαίτερα εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος. Σύμφωνα με τους αριθμούς μας, είχαμε άνω των 600 συμμετεχόντων, κάποιες στιγμές τουλάχιστον, Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και δείχνει το ενδιαφέρον που έχει ο κόσμος για τα θέματα αυτά και θα πρέπει το ενδιαφέρον αυτό να προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε στο μέλλον. Ξέρω ότι ο Πολωνός υπουργό είναι εδώ και διαρωτώ με. Είναι δύσκολο να σας βλέπω εκεί που κάθεστε, κρύβεστε από μένα. Αλλά θα ήθελα να σας προσκαλέσω αν θέλετε ε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να μας μεταφέρετε τις απόψεις σας και να σχολιάσετε λίγο το φόρουμ το οποίο θα διεξαχθεί σε ένα χρόνο στη χώρα σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Βελγική Προεδρία για την οργάνωση για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες αυτού του φόρουμ για την ενιαία αγορά. Αναγνωρίζουμε έτσι τη σημασία της ενιαίας αγοράς για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Αυτό φαίνεται και στην πρόταση του Μόντι και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και δύο εβδομάδες για την ενιαία πράξη. Η πρωτοβουλία αυτή του Φόρουμ προήλθε φυσικά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως είδαμε σήμερα την χάνει ισχυρή στήριξη. Τέθηκαν πολύ σημαντικά θέματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σήμερα για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην οικονομία θα πρέπει να, υπάρξει να σωστή διακυβέρνηση και φιλόδοξη διακυβέρνηση της οικονομικής ε, δραστηριότητας στην Ευρώπη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το φόρουμ αυτό θα πρέπει να γίνεται ετήσια, σε ετήσια βάση, θα πρέπει ε, να γίνεται κατέτος στην ε, χώρα που έχει την Προεδρία και θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους στο επόμενο φόρουμ για την ενιαία αγορά που θα γίνει στην Πολωνία το φθινόπωρο του 2011 κατά τη διάρκεια της πρώτης πολωνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στόχος μας είναι να φέρουμε σε επαφή εκπροσώπους επιχειρήσεων, καταναλωτών, εκπροσώπους των κρατών μελών και να δημιουργήσουμε μια σημαντική πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και ε, χρηστών ή μάλλον βέλτιστων πρακτικών. Να υπάρξει σωστή ενημέρωση των πολιτών, των δικαιωμάτων των πολιτών και των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων. Η χρονιά που μεσολαβεί ε, σημειώνει πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την ενιαία αγορά, προκλήσεις για το 2020, η έκθεση για τις προκλήσεις αυτές, θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή βάση για τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες και αυτό θα γίνει και στην Πολωνία. Ελπίζω ότι με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής θα κάνουμε και μια προπαρασκευαστική συνάντηση για να γιορτάσουμε ε, το 2012 τα 20 γενέθλια της ενίας αγοράς. Ελπίζω να σας δούμε όλους λοιπόν στο δεύτερο φόρουμ για την ενιαία αγορά στην Πολωνία σε ένα χρόνο από σήμερα. Uh, uh, uh, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ που πήρατε το λόγο, πολύ ενθαρρυντικά τα λόγια σας. Προτού ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την ομάδα μου που βρίσκεται εδώ πέρα στο πάνελ, τον Λουίς Γκρέχα και τον κύριο Μπουζόη, που ανέλαβαν το συντονισμό των ε, διαφορετικών πάνελ, καθώς επίσης και τη σημαντική δουλειά που έχουν κάνει ως για πολύ σημαντικές εκθέσεις. Όπως βλέπετε πρόκειται για μια πραγματική εργασία ομάδος, μια ομαδική εργασία. Υπάρχουν πολλά μέλη από την Επιτροπή ε, Εσωτερικής Αγοράς που έχουν συνεργαστεί επικοδομητικά δεν σημαίνει αυτό ότι συμφωνούμε για τα πάντα. Συμφωνούμε όμως ότι θέλουμε να ακολουθήσει η νέα αγορά μια ξεκάθαρη κατεύθυνση προκειμένου να δημιουργήσει πραγματικά ωφέλη για τους καταναλωτές, όπως είπε η κυρία Κόιενς, αλλά και για τους πολίτες. Δηλαδή να δοθεί δυνατότητα στους πολίτες να μετακινούνται πιο εύκολα, να γνωρίζουν τα προσόντα τους, να είναι σε θέση να αν λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να καινοτομούν. Και όπως είπε και ο Μάριο Μόντι, δημιουργείται μια γανάκτηση σε πολλούς από εμά το ότι ε, δεν έχουμε καλύψει όλο αυτό το έδαφος το οποίο θα έπρεπε να έχουμε καλύψει. Είναι σημαντικό τουλάχιστον ότι καταφέρουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε κάποιες δεσμεύσεις πλέον από τα κράτη-μέλη με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες. Και το πρώτο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη θα σεβαστούν, θα τηρήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ καλύτερο να έχουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα από το να έχουμε κάτι το οποίο δεν θα τηρήσουν τελικά τα κράτη-μέλη, κάτι το πιο φιλόδοξο, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί στην πράξη. Θέλουμε όχι φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους θα προτιμούσα να περάσω περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσω τη δέσμευση από τα κράτη-μέλη από το να αφιερώσω χρόνο στην κατάρτιση ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου σχεδίου που δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί όμως. Αφού ευχαρίστησα λοιπόν τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία της Επιτροπής, η οποία εργάστηκε πάρα πολύ για τη διοργάνωση της σημερινής συζήτησης και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εμαντέλε και Πάμελα Ντόνσορ, καθώς επίσης και όλη την ομάδα τους που ήταν εδώ και που ε, Καταρχά, κατέβαλαν πάρα πολλέ προσπάθειε για την ίδια την εκπόνηση τη πράξη για την ενή αγορά, αλλά και συνέβαλαν πάρα πολύ στην ε, πρακτική διοργάνωση τη σημερινή συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Να ευχαριστήσω όμω και το Συμβούλιο και τους εκπροσώπους Συμβουλίου. Οι εκπροσώποι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Είδατε ότι είχαμε εκπροσώπηση σε υπουργικό επίπεδο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την υφιστάμενη όσο και τη μελλοντική, τις μελλοντικές προεδρίες. Επίσης πρέπει να σας πω ότι θα είδατε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα. Έφτασε και ένα νέο σήμερα, αυτό το φυλάδιο το οποίο κρατάω στα χέρια μου. Έχουμε επίσης και το ενημερωτικό φυλάδιο της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς. Μπορείτε να γραφτείτε ηλεκτρονικά. Κατά αυτόν τον τρόπο θα λαμβάνετε το ενημερωτικό μας φυλάδιο σε τακτική βάση. Βλέπετε επίσης τα ονόματά μας καθώς επίσης και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο πίσω μέρος της, του φυλαδίου αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση ο πρόεδρο και όλου αυτού που μα παρακολουθούν από το διαδίκτυο και εύχομαι σε όλους, σα, είστε βρίσκεστε κάπου στον κυβερνοχώρο ή στι Βρυξέλλες ένα πολύ καλό βράδυ. Σα ευχαριστώ.